Mes chers collègues, euh, je vous propose de démarrer notre euh, réunion extraordinaire de ce matin. Αγαπητοί συνάδελφοι, σα προτείνω να αρχίσουμε την έκτακτη συνεδρίαση. Θα έρθει η Έλγα Στέβεν, περιμένω λίγο. Σίγουρα θα έχει ε, μπλοκαριστεί στην κίνηση. Σε πέντε λεπτά ακούω. Εντάξει, πέντε λεπτά, αλλά να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας και θα έρθει η Καστίβερ. Καλημέρα σε όλους και σας ευχαριστώ όλους σας για την παρουσία σας εδώ την τελευταία μέρα της συνόδου μας. Λοιπόν, πάμε μέσω στην ημερήσια διάταξη τη σημερινή που είναι έτσι κάπως πιο ιδιαίτερη και να αρχίσουμε τον κλασικό τρόπο. Σημείο πρώτο, έγκριση της ημερησίας διάταξης. Έχετε αντιρρήσεις? Αν δεν διαφωνεί κανεί, θεωρείται εγκεκριμένη ημερήσια διάταξη. Και περνάμε στο σημείο 2, ανακοινώσει τη Προεδρία. Την περασμένη φορά που συνεδριάσαμε στις 19 Ιουνίου, οι συντονιστές συμφώνησαν ε, σε διάφορα σημεία. Πρώτα απ' όλα να προσκαλέσουμε τον κύριο Γκίντερ Ότιγκερ, ε, τον ε, Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τον προπολογισμό και τους ανθρωπίνους ε, πόρους και τον κύριο Ζίλντε Κέρκοφ που είναι συντονιστής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας την άλλη εβδομάδα που έχουμε συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Και ευχαριστώ τη Γραμματεία για την αποτελεσματικότητά της όταν και τι προσπάθειε που έκανε για το συντονισμό και τη συνεργασία. Επίση, οι συντονιστέ αποφάσισαν να γίνει δημόσια ακρόαση για την προστασία των κρισίμων υποδομών και των δημοσίων χώρων την άλλη εβδομάδα στι 12 Ιουλίου στι Βρυξέλλε. Και επίση αποφάσισαν να καλέσουν τον Σερ Τζούλιαν Κίνγκ, Επίτροπο Αρμόδιο για την Ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην έκτακτη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα ΤΕΡ στο Στρασβούργο στι 13 Σεπτεμβρίου. Με το καλό. Επίσης, ε, αποστολή στην Αβέρσα στο Λιμένα έχει εγκριθεί το πρόγραμμα ε, καθώς επίσης και ο τρόπος κατανομής ε, των θέσεων σε αυτή την αποστολή η οποία αποστολή θα γίνει την άλλη εβδομάδα επίσης στις 12 του μηνός Ιουλίου Βρυξέλλες Αμβέρσα εντάξει αποστολή θα βρείτε τις λεπτομέρειες μπορεί να τις έχετε ήδη λάβει αυτά ως προς τις ανακοινώσεις και αν συμφωνείτε να περάσουμε στο βασικό θέμα της σημερινής διάταξης που αφορά τις συστάσεις και προτάσεις της ειδική μας Επιτροπής για την Τρομοκρατία ε, με το σχέδιο έκθεση το οποίο θα εξτάσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε την έκθεση από χτες τουλάχιστον σε όλες τις γλώσσες. Euh, donc été euh, euh, envoyé, je pense, à tous les membres. Ε, σε όλα τα μέλη. Και σας προτείνω, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, να δώσουμε μέσω στο λόγο στις δύο συνεισηγήτριές μας, που είναι η κυρία Μόνικα Χόλμαια και η κυρία Χέλγα Στέβενς, για να μας παρουσιάσουν την έκθεσή τους. Εντάξει, θα έρθει η Χέλγα κάποια στιγμή. Να αρχίσουμε με τη Μόνικα και βλέπουμε. Παρακαλώ. Θα πρότεινα το εξή να ακούσουμε πρώτα τις δύο εισηγήτριές μας και μετά τους σκιώδεις εισηγητές Θα έχουμε πρώτα την κυρία Κινίτσι για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η Μάιτα Παγάσα Ορτοντούα από τους φιλελευθέρους, η κυρία Εύα από την ομάδα των Πρασίνων, η κυρία Βερζιά από την ΚΟΕ και ε, ο κύριος Δομινίκ Μαχτάν, τον οποίο δεν βλέπω, από την ομάδα ΙΕΝΕΦ. Στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στο γενικό, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Αρμόδιας Ελληνικής Διεύθυνσης για να μας πει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Και στη συνέχεια, στον υπόλοιπο χρόνο που θα μας έχει απομείνει, θα κάνουμε ερωτήσεις και απαντήσεις αναλόγως ό,τι προλάβουμε με τη διαδικασία CATS Αυτά. Και αν συμφωνείτε όλοι, θα δώσω αμέσως το λόγο στη Μόνικα Χόλμα ε, να μας κάνει την παρουσίασή της. Παρακαλώ, Μόνικα. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ορισμένοι έχουν δυσκολίες να μπουν στο κοινοβούλιο. Ήμουν 20 λεπτά έξω από την πύλη και δεν με αφήνανε να μπω. Καμία περίπτωση καμία πιθανότητα. Ελπίζω και η Χέλγα να μην έχει κολλήσει έτσι. Ήταν μπλοκαρισμένη όλη η παράδρομη και δεν μπορούσε να περάσει κανείς να φτάσει στο κοινοβούλιο. Μπορεί και η Χέλγα Στίβενς κάπου εκεί να έχει κολλήσει. Ε, ελπίζω να προλάβει, να μπορέσει να έρθει. Λοιπόν, ε, καταρχάς θέλω να πω ότι δουλέψαμε όλους αυτούς τους μήνες πολύ εντατικά και φτάσαμε στη σημερινή τελική έκθεση. Και εγώ προσπάθησα ως εισηγήτρια να συμπεριλάβω όλα αυτά ε, που είχαμε αποκομίσει από αποστολές, από συζητήσεις με τα κρατη με εμπειρογνώμονες. Είναι τεράστιο το φάσμα και ε, ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων. Καταφέραμε ή προσπαθήσαμε τουλάχιστον κάπως να τα ε, συνεφέρουμε αυτά και να τα συμμαζέψουμε όλοι οι συνάδελφοι που έχουν εργαστεί στην Επιτροπή αυτή έχουν καταλάβει πόσο ευρύ είναι το θέμα ε, και πόσο πολυεπίπεδα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Δεν είναι καθόλου απλό έτσι ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί στην δράση μας και στην καταπολέμηση. Γεια σου Χέλγα! Ορίστε, τα κατάφερε και η Χέλγα. Ε, ε, με τους και οδησηγητές συνεργαστήκαμε πολύ αγαστά και θέλω να τους ευχαριστήσω επίσης, αλλά και τους συντονιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καταπληκτική συνεργασία και τη γραμματεία. Γιατί χρόνο πολύ δεν είχαμε, ήταν πολύ περιορισμένος ο χρόνος και θα πρέπει να το πούμε και αυτό αγαπητή κυρία Πρόεδρε, γιατί μόλις εννέα μήνες για να δουλέψουμε. και να καλύψουμε όλο αυτό το φάσμα δεν είναι καθόλου εύκολο. Ευχαριστώ και την Πρόεδρο για την κατανόησή της. Και όποτε θέλαμε να καλέσουμε κάποιον εμπειρογνώμονα και τα λοιπά, πάντα ήταν στη διάθεσή μας. Ε, απόλυτη υποστήριξη και η Πρόεδρος και όλο το επιτελείο. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι με τη Χέλγα ε, μοιραστήκαμε λίγο τα θέματα και εγώ ασχολήθηκα κυρίως με την ε, αξιολόγηση της απειλής, αυτό το threat assessment ε, και απευθυνθήκαμε σε όλες τις αρχές ασφαλείας, κυβερνήσεις, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες κλπ. Για να δούμε εάν εκτός αυτών που βλέπουμε έτσι να κυκλοφορούν δημόσια, αν υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι και απειλές παγκοσμίω. Πέρα από τον ΤΑΕΣ, το ISIS δηλαδή και την Αλκάιντα, υπάρχουν έτσι μεγάλες απειλές αυτή τη στιγμή από πλευρά των δημοκρατικών οργανώσεων ή άλλων ομάδων που μπορεί να μην έχουμε καν αντιληφθεί και υπήρξε σαφής απάντηση ότι όχι, υπάρχουν μεμονωμένα επεισόδια, ακροδεξιοί, εξτρεμιστές, ακροαριστεροί, αυτονομιστές κτλ. Αλλά δεν υπάρχει παγκόσμια, ε, ευρωπαϊκή μεγάλη οργάνωση που να συνιστά τόσο μεγάλη τρομοκρατική απειλή όπως αυτές που γνωρίζουμε ή να εξελίσσεται προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά με την Ισλαμιστική τρομοκρατία ε, αυξάνονται και οι απειλές ε, στα άκρα του πολιτικού φάσματος. Και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα στεναρά. Πολύ βασικό αυτό. Επίσης, ασχοληθήκαμε και με το εξής τα κράτη-μέλη έχουν νομοθεσία, έχουν νομοθετικά μέτρα και πώς τα εφαρμόζουν. Και ε, εδώ έχουμε πάντα ε, ελλείμματα, προβλήματα, διαφορετική αντίληψη για την πραγματικότητα, ε, καμιά φορά διστακτικότητα. Πού οφείλεται αυτό. Υπάρχουν κάποιοι κρατημέλη που οφειλεται αυτο υπαρχουν καποιοι μελη που μάλλον που θεωρούν ότι δεν τους αφορά η τρομοκρατία και δεν βάζουν ε, στοιχεία στις τράπεζες δεδομένων. Ή κάποιες χώρες που δεν έχουν ε, εμπειρία με την τρομοκρατία εφαρμόζουν με πολύ στοιχειώδη και βασικό τρόπο την νομοθεσία. Είναι πιο διστακτικά και απρόθυμα. Εμείς θέλουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο να εφαρμόζεται σωστά, με συνέπεια και εάν ε, κάποιος αντιδρά και αδρανεί ή εσκεμμένα δεν την εφαρμόζει θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το επιβάλλει γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια τέτοια κουρελού από μέτρα. Ε, αυτό είναι πρόβλημα και στη συνεργασία. Επίσης ασχολήθηκα με το θέμα της ανταλλαγής ε, πληροφοριών και μαζί σας και με τη Χέλγα και διαπιστώνουμε ότι και εκεί είναι πολύ διαφορετική η τακτική και η συμπεριφορά των κρατών μέλων. εκεί έχουμε ακόμα και τεχνικά εμπόδια και νομικά αλλά και αντικειμενικά προβλήματα. Τι εννοώ αντικειμενικά πρόβλημα σε ανθρωπίνους πόρους και οικονομικούς πόρους ή ανεπαρκώς ε, καταρτισμένο προσωπικό. Στα κράτη-μέλη τι γίνεται. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και τα πρότυπα και τα στάνταρ δηλαδή, αλλά και τα κέντρα βάρους και οι προτεραιότητες των κρατών μελών. Επίσης, στην ανταλλαγή των πληροφοριών είχαμε και πολύ συγκεκριμένα και τεχνικά που μάθαμε και νομικά προβλήματα. Και συχνά κάναμε συζητήσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Όταν, για παράδειγμα, τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετική νομοθεσία ε, και πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες ε, με άλλα κράτη-μέλη. Ας πούμε, πόσο κρατάμε ε, τα δεδομένα. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι τεράστιο το φάσμα των μέτρων που έχουν τα κράτη-μέλη και των νομοθεσιών. Πώς θα συνεργαστούν για την ανταλλαγή προφοριών όταν ισχύει όλο αυτό το αλαλούμ και ε, με πολύ διαφορετικό τρόπο αντιλαμβάνονται τα κράτη-μέλη καν αυτή την προσπάθεια. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Είμαι στη διάθεσή σας να εξηγήσω σε κάθε σημείο τι εννοώ. Είχαμε πάντα συζητήσεις γιατί δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες ας πούμε ή δεδομένα και στοιχεία τα κράτη-μέλη τα οποία κανονικά αυτά πρέπει αυτόματα να ανταλλάσσονται. Υπάρχει μια πρόταση να γίνει ακριβώς αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών εκτός εάν υπάρχει λόγος ξέρω εγώ, κρατικής ασφάλειας και τα κράτη-μέλη ε, το σταματάνε γιατί δεν, δεν έχουν έγκυρα στοιχεία υπάρχει αυτό που λένε information exchange by default. Είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτής της πρότασης, γιατί αν έχουμε ευρωπαϊκό δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο ορισμένα πράγματα και ορισμένες ε, πληροφορίες συγγνώμη, ε, ανταλλάσσονται και διαβιβάζονται υποχρεωτικά, δια νόμου δηλαδή είσαι υποχρεωμένος, τότε θα πρέπει αυτό να γίνεται αυτόματα. Και να γίνεται όμως. Επίσης, και η Χέλγα Στέβενς και εγώ χαιρόμαστε για τις προτάσεις ε, διαλειτουργικότητας για τα κεντρικά συστήματα προφορίας ένα πρώτο βήμα είναι αυτό και σημαντικό αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις εθνικές τράπεζες δεδομένων και ποια σχέση θα έχουν αυτά τα δύο και ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν στο μέλλον και έχουμε μια παράκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το δει αυτό εντατικά γιατί πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την κουρελού και τον κατακαιρματισμό που έχουν τα κρατη Έχουμε ακούσει τέτοια πράγματα από τις αρχές ασφαλείας, από εισαγγελείς, από δικαστές, ότι ε, όταν ε, συγκεντρώνουν κάποιες πληροφορίες, τότε και μόνο τότε έχουν κάποια εικόνα. Δηλαδή μπορεί με μονομένες ε, πληροφορίες να φαίνονται ανώδυνες, αλλά εάν τις συνδυάσεις με κάποιες άλλες, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ολόκληρο δίκτυο από πίσω. Δηλαδή είναι σημαντικό οι πληροφορίες αυτές αυτές να ανταλλάσσονται, να μην θεωρεί κάποιος ότι είναι ασήμαντη και να μην τη διαβιβάζει. Και η Ευρωπόλ θα πρέπει να γίνει ένα hub πληροφόρησης ή ανταλλαγής πληροφοριών καλύτερα, έτσι ώστε να συντονίζει και να είναι ένα κεντρικό σημείο ε, ε, διαβίβασης πληροφοριών με τους γνωστούς κανόνες διαφάνειας και προστασίας δεδομένων που από κοινού έχουμε θεσπίσει. Μετά ασχοληθήκαμε με τα θέματα της ριζοσπαστικοποίησης. Χωρίς να μπω τώρα σε όλα τα μέτρα σε λεπτομέρειες, σύμφωνα με την άποψη της Χέλγα και τη δική μου, και ελπίζω να συμφωνείτε με την κατεύθυνση, υπάρχει ένα ολόκληρο συμβίλημα ε, μέτρων ε, που είναι από την ένταξη στην κοινωνία μέχρι κατασταλτικά μέτρα. εάν κάποιος ε, κηρύσει το μίσος ας πούμε και προτρέπει τον κόσμο να βιάζει γυναίκες, σε κάτι πρέπει να του συμβεί. Δεν μπορεί να καταργεί το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ο καθένας και να κηρύσει το μίσος και ε, αυτά να συμβαίνουν ατιμωρητή και μάλιστα ε, και να προσπαθεί να το προβάλλει και ως δόγμα πίστης σε μια μουσουλμανική κοινότητα αυτό. Επίσης ασχοληθήκαμε με τη χρηματοδότηση, την έξωθεν και τι διαπιστώσαμε στην ανάλυση αυτή, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιρροή των ουαχαμπιτών και οικονομικά προσπαθούν να το προωθήσουν, ε, χρηματοδοτούν πολύ ακραίες ε, φονταμενταλιστές ε, οργανώσεις, οικογένειες συγκεκριμένες από κάποιες τρίτες χώρες χρηματοδοτούν αυτούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διάφορα Ινστιτούτα και θεσμούς εγνωσμένου κύρους. Αν θέλετε πληροφορίε μπορούμε να σας τα δώσουμε τα στοιχεία από πανεπιστήμια που μας έχουν στείλει. Δεν μπορέσαμε να τα επεξεργαστούμε όλα, μόνο έτσι κάπως ακροθυγός γιατί φτάνει μέχρι και σε χρηματοδότηση πανεπιστημίων, ε, κατάρτισης, ε, χρηματοδοτούν ε, θεολογικές σχολές που εκπαιδεύουν οι μάμιδε, ακόμα και τεμένοι. Ε, με πολύ ακραίες ερμηνείες του Κορανίου. Υπάρχει κινηματογραφικό υλικό, υπάρχει υποστήριξη ε, όλης αυτής της φιλοσοφίας, της ριζοσπαστικής ε, από το διαδίκτυο. Αυτό δεν είναι ακόμα προπαγάνδα υπέρ της τρομοκρατίας, αλλά είναι στην κρίζα ζώνη της παραβίασης του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, χωρίς ακόμα να μπαίνει σε αξιόπινες πράξεις, ας πούμε, σε προτροπή για τρομοκρατία. Είναι στον προθάλαμο της τρομοκρατίας όλα αυτά. Πολύ προβληματικός τρόπος χρηματοδότησης και προώθησης αυτών των ιδεών. Τελευταίο. Τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Στην Ισπανία μου έκανε μεγάλη εντύπωση η επίσκεψη. Δεν ξέρω οι συνάδελφοι πώς το ένιωσαν αυτό, γιατί έχουν μακρά εμπειρία και πολύ επώδυνη δυστυχώς, και γνωρίζουν τι γίνεται και πώς ε, ε, μεταχειρίζεται τα θύματα και τι κάνεις και το καθεστώς του θύματος έχει προχωρήσει πολύ και είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι σε άλλα κράτη-μέλη, σε πολλά έχουν δικές τους οργανώσεις, εκπρόσωποι των θυμάτων, μέχρι και επιστημονικό επίπεδο είναι αναγνωρισμένοι και συμμετέχουν σε όλα τα μέτρα που λαμβάνονται. Είναι συνομιλητής οι οργανώσεις των οικογενειών των θυμάτων. Θα πρέπει και εμείς να το επιδιώξουμε αυτό, διότι τα θύματα της τρομοκρατίας δεν θα πρέπει να γίνονται διπλά θύματα, κάθε φορά να τους θεωρούμε θύματα και όχι συμμετέχοντες σε μια διαδικασία ε, καταπολέμησης όλων αυτών. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε να μην γίνονται οι άνθρωποι αυτοί επέτες, ε, να μην ζητιανεύουν ε, νομικά θέματα, κοινωνικά θέματα, να μην ε, ζητιανεύουν καν να εισακουστούν. Θα πρέπει να φροντίσουμε να συμμετέχουν από την αρχή τα θύματα και οι οργανώσεις τους να είναι γνήσιοι αυθεντικοί συνομιλητές και για αυτό που του συνέβη. Να παίρνουν πλήρη αποζημίωση και το κράτος να είναι αρμόδιο και υπεύθυνο. Γιατί η τρομοκρατία δεν πλήττει τους ανθρώπους γιατί έχουν κάνει κάτι κακό ή γιατί έχουν τσακωθεί με κάποιον ή έχουν θυμώσει. Είναι ε, μια επίθεση ε, κατά του κράτους, κατά των αξιών μας και, και την πάτησαν γιατί ήταν τυχαία εκεί και έγιναν θύματα. Ε, άρα το κράτος θα πρέπει να αναλαμβάνει να αποζημιώνει τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Επίσης, η Κατερίνα Κινίτσι ε, ζήτησε να υπάρξει ένα ξεχωριστό κλάστερ ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην έκθεση με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά κύριο λόγο θα το δούμε πώς θα γίνει, πώς θέλετε να το βάλουμε αυτό το κεφάλαιο, να συνεργαστούμε. Απλώς θέλουμε να πούμε ότι για μας ισχύει όλος ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων τελεία, στο εκαίρεο. και κάθε σημείο ξεχωριστά. Δεν ήθελα τώρα να απομονώσω κάποια σημεία ή κάποια δικαιώματα και να αφήσω στην άκρη κάποια άλλα. Αλλά ε, ο τραυματισμός ε, και ο σωματικός και ο ψυχο, ψυχικός είναι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί στη ζωή σου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χέλγα. Είχαμε καταπληκτική συνεργασία και θέλω να σταματήσω για να συνεχίσει και η Χέλγα, αν μας το επιτρέπει, πρόεδρος. Σα ευχαριστούμε πολύ, Μόνικα. σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση αυτή και θα δώσω κατευθείαν το λόγο στη Έλγα Στίβεν, η οποία έχει καταφτάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα σας και το συγγνώμη για την ε, καθυστέρηση, γιατί πήρε το λόγο στην Ολομέλεια σε ό,τι αφορά την πολιτική συμμετοχή των ατομών με αναπηρία το οποίο είναι ασφαλώς και δικό μου φάκελος. Πρώτο λοιπόν ξεκινήσω, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω την συνάδελφό μου τη Μόνικα για την καλή συνεργασία. Είναι πραγματικά χαρά μου το γεγονό ότι συνεμονούμαστε τόσο καλά σε επίπεδο πολιτικών ομάδων επί του περιεχομένου. Η καταπολέμηση τη τρομοκρατία ε, περνάει πέρα από τα σύνορα των πολιτικών ομάδων και ελπίζω ότι η σημερινή συζήτηση θα είναι επικοδομητική και θα είναι και στάση μας επικοδομητική του επόμενους μήνες προκειμένου να καταρτήσουμε ένα κείμενο οράματος το οποίο θα είναι αποδεκτό για όλες τις πολιτικές ομάδες και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα άλλα μέλη της Επιτροπής για τις ε, παρεμβάσεις σας ε, κατά τη διάρκεια της ανακροάσεων των συνεδριάσεων της Επιτροπής ε, και στις αποστολές. Να ευχαριστήσω επίσης για την υπομονή σας. Η κατάρτιση λοιπόν του σχεδίου έκθεσης ε, πήρε χρόνο. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε την έκθεση που παρουσιάζει το, την προσέγγιση των συναδέλφων μου και της αντιπροσωπείας μου του ΕΝΒΑ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας λοιπόν να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις με προστιθέμενη αξία. Σε τελική ανάλυση θεωρώ ότι το κείμενο είναι πολύ ζωντανό που αποτυπώνει την ευρεία εντολή που έχει αυτή η προσωρινή μας επιτροπή. Εγώ λοιπόν άκουσα και τις ε, βασικές ε, ε, προτάσεις της Μόνικα και θα θέλαμε να ακούσουμε τώρα και ποιες είναι οι δικές σας οι απόψεις από αυτών των προτάσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιες συστάσεις τις συμπεριλάβαμε από τις εκθέσεις που έχουν ήδη εγκριθεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάποια θέματα δεν ήταν απαραίτητο να επενεφεύρουμε τον τροχό. Για παράδειγμα, το πιστοποιητικό για τον εντοπισμό τέχνης προκειμένου κλοπημαία από περιοχές συγκρούσεων να μην χρηματοδοτούν έμεσα ή άμεσα τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό λοιπόν ήδη έχει λάβει υπόψη τις τοποθετήσεις όλων των πολιτικών ομάδων και η έρευνα και οι συστάσεις ε, της Βελγικής Επιτροπής ε, του Κοινοβουλίου, του Βελγικού Κοινοβουλίου συμπεριλήφθησαν στη συζήτηση. Θα διαβάσετε λοιπόν κάποια συστάσεις σε ό,τι αφορά την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων. Η περιοχή Σέγγεν χωρίς εσωτερικά σύνορα μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει μόνον εφόσον τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προστατευτούν αποτελεσματικά. Και κάποιες από τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις ε, αποκάλυψαν μεγάλες ελλείψεις ε, στην ευρωπαϊκή πολιτική για την ταχύτητα των εξωτερικών συνόρων. Για παράδειγμα, η επίθεση στο τρένο τα Θαλής ε, και στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες αποκάλυψαν ότι οι εγκέφαλοι πίσω από τις τρομοκρατικές αυτές οργανώσεις είχαν μπει στην Ευρώπη μέσω παράνομων μεταναστευτικών νερών, τον Ιούλιο, Αύγουστο και Οκτώβριο του 2015 μέσω της Ελλάδας. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν οι σωστές ε, προϋποθέσεις στα εξωτερικά σύνορα για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, να υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, βιομετρικών ελέγχων, να υπάρχει διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων και να χρησιμοποιούνται όλα τα δεδομένα και τα PNR για να εντοπίζονται ενδεχόμενοι τρομοκράτες που μπαίνουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωρίζουμε ότι η UNAFOR με την ε, επιχείρηση Σόφια αποτελεί την μεγαλύτερη τρέχουσα επιχείρηση στη Μεσόγειο και διαθέτει, ε, διαθέτει μέτρα και μέσα για να καταπολεμήσει την τρομοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε να προσαρμοστεί η εντολή της επιχείρησης Σόφια και να επεκταθεί, να συμπεριλάβει και την Τινησία για να καταπολεμήσει τις χώρες ε, υποδοχής όπως ονομάζονται στη Σαρδινία και το καθεξής. Και έτσι λοιπόν εξετάζουμε την ε, ενδεχόμενη πρόσβαση της Σοφία και στα χωρικά ύδατα της Λιβύης για να ελέγχονται τα σκάφη και εκεί. Συνάδελφοι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονό ότι και η Γυροπόλ συμπεριλαμβάνεται στην επιχειρήση Καλάν Φίνιξ στην ε, Ιορδανία. Γιατί έχουμε πληροφορίες ότι μαζεύονται δυνάμει στη Λιβύη και αλλού. Αυτά μα λέει η Γυροπόλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα δεδομένα να μπουν και σε βάση δεδομένων προκειμένου να τα έχουν στη διάθεσή τους και οι συνεργοφύλακε κατά τη διάρκεια του ελέγχου των ατόμων που θέλουν να εισέλθουν στην Ένωση. Επίση, είναι σημαντικό να υπάρξει εναρμόνεση των ε, οικονομικών υπηρεσιών των εθνικών κρατών μελών, γιατί δεν υπάρχει τέτοια εναρμόνεση και δεν γίνεται σωστή ανταλλαγή δεδομένων. Το FEU αυτή η πλατφόρμα θα πρέπει να διευρυνθεί προκειμένου να είναι πιο εύκολη η διμερή ανταλλαγή και δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρχουν σωστά μέσα για την ε, καταπολέμηση της μακρο μεγάλης κλίμακας χρηματοδότησης των δημοκρατικών οργανώσεων και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε πλήρως ε, τις οικονομικές πληροφορίες για να υπάρχει σωστή πρόληψη προκειμένου και η αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας και οι μυστικές υπηρεσίες να μπορούν να δράσουν πιο πολύ προληπτικά. Η δυνατότητα εντοπισμού των τρομοκρατικών οργανώσεων και καταγραφής ε, των τρομοκρατικών οργανώσεων δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εθνικές ε, υπηρεσίες μπορούν να υποβάλουν λοιπόν μια τέτοια ένα τέτοιο αίτημα στο FTP και το σύστημα, αυτό το σύστημα ανταλλαγής ε, πληροφοριών. Οι συναλλαγές ΕΠΑ όμως εξαιρούνται. Ζητούμε κατεπηγόντω να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σύστημα FTP προκειμένου και οι συναλλαγέ ΕΠΑ να παρακολουθούνται. Το πώ θα δημορφωθεί ακριβώ το σύστημα το συζητάμε. Υπάρχουν διάφορε δυνατότητε. Ένα υβριδικό σύστημα ενδεχομένω ενδεχομένω μια κεντρική υπηρεσία η οποία θα είναι σε επαφή με τι εθνικέ ε, υπηρεσίε για την ενίσχυση του δικτύου FTE. Ζητάμε λοιπόν να αναφερθεί το 214, το 2014 προκειμένου οι κρίσιμες υποδομές να προσαρμοστούν βάσει ανάλυση των συστημάτων σε ό,τι αφορά τις ε, διασυνοριακές υπηρεσίες, όχι βάσει τομεακής προσέγγισης. Ε, στη νέα λοιπόν οδηγία θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση καταγραφής κάθε περιστατικό που θα έχει να κάνει με τις κρίσιμες υποδομές και στο πλαίσιο των stress test. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν προσαρμογή των σημείων επαφής και προϋποθέσεις ε, ποιότητας και ασφάλειας σε ό,τι αφορά τη συνέχεια των επιχειρήσεων σε περίπτωση επιθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαθέσει μέσα από πανευρωπαϊκά συστήματα όπως Γαλλιαίο και Eurocontrol ως ευρωπαϊκές ε, κρίσιμες υποδομές το 2015 και το 2016. Σε 40% των ε, ε, τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά και παρά το γεγονός ότι ο κανονισμός 98-2013 προβλέπει να παρέχονται σε ιδιώτε, σε ουσίε σε περιορισμένες ποσότητες και να καταγράφονται οι συναλλαγές αυτές. Και ο λόγος είναι ότι οι οι τρομοκράτε μπορούν να εξακολουθούν να έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν τα εκρηκτικά αυτά online, στο διαδίκτυο και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν δυνατότητα να εφαρμόζουν διάφορα συστήματα. Άρα ζητάμε να υπάρχει πιο αυστηρή παρακολούθηση και εποπτεία των αγορών στο διαδίκτυο για να προσαρμοστούν επίσης ε, πιο αυστηρά κριτήρια σε ό,τι αφορά τα τελωνία προκειμένου να υπάρχει καλύτερο συντοπισμό τελικά αυτών των ε, ουσιών. Χρειάζονται λοιπόν πρακτικά μέτρα και είναι θέμα ζωή ή θανάτου. Άρα χρειαζόμαστε παρακολούθηση των online πλατφορμών για ουσίες ε, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή εκρηκτικών ε, και να υπάρχει σωστή, σωστή συντοπισμό, σωστό συντοπισμό των ουσίων αυτών. Τέλος, θα πρέπει να βελτιωθούν οι φυστάμενες δομές και σε εθνικό επίπεδο όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, συστήσουν ένα κέντρο αντιμετώπιση κρίσεων για εθνικέ κρίσει και για να δημιουργηθεί έτσι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο τέτοιων υπηρεσιών. Όντω, χρειάζεται κάθε κράτο μέλο να έχει ένα κέντρο συντονισμού και να συνεργάζονται με την Ευρώπη των 28 χρησιμοποιώντας τις υποδομές EPCR σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του Ιουνίου του 2017 σε ό,τι αφορά την γενική ευαισθητοποίηση των πολιτών και τις αντιλήψεις των πολιτών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, το αίσθημα ασφάλειας, 92% ε, των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι οι εθνικές υπηρεσίες θα πρέπει να μοιράζονται υπηρεσίες, ε, πληροφορίες με τις υπηρεσίες άλλων κρατών μελών προκειμένου να καταπολεμηθεί καλύτερα το έγκλημα και η τρομοκρατία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια νέα νοοτροπία και θα πρέπει να προωθηθεί αυτή η νοοτροπία για την ε, κοινή χρήση των πληροφοριών και μόνο σε ιδιαίτερε περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει εξαίρεση από την υποχρέωση και είναι αυτονόητο ότι συμφωνώ και με τι συστάσει τις οποίες έκανε πριν από λίγο η συνάδελφός μου η Αυστριακή κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα να κλείσει 7 τζαμιά και να ε, εκδιώξει 60, να απελάσει 60 ημάμιδες ε, που κάναν προπαγάνδα για το πολιτικό Ισλάμ. Το υποστηρίζω αυτό απόλυτα, γιατί οι ημάμιδες που δεν τηρούν τις ευρωπαϊκές αξίες και υποκινούν για τρομοκρατία, προς τρομοκρατία, δεν έχουν ε, θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να τονίσω ότι ένα κράτο δικαίου το οποίο λειτουργεί σωστά είναι το κλειδί για την καταπολέμηση της τρομοκρατία. Όχι μόνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, όπως και το δικαίωμα τη ιδιωτική σφαίρας, αλλά γιατί χρειάζεται σωστή δικαιοσύνη, χωστό σύστημα δικαιοσύνη για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία τι γίνεται με το ποινικό μητρό. Η αστυνομία κάνει αυτά που τη αναλογούν. Θα πρέπει και η δικαιοσύνη λοιπόν να κάνει αυτά που τη αναλογούν. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή ε, ποινικοποίηση τέτοιων πράξεων. Γιατί αν υπάρχει γενικώ αίσθηση ασυνδοσία, θα υπάρχει και ανεξέλεγκτη ριζοσπαστικοποίηση και θα στρεφόνται κατά των πολιτών. Αυτά. Και Προσβλέπω και ανυπομονώ να ακούσω τι παρεμβάσει σα και τι παρατηρήσει σα. Η πόρτα του γραφείου μου είναι μονίμω ανοιχτή για να ακούσω τι έχετε να μου πείτε και θα ήθελα εκ νέου να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο τη Μόνικα αλλά και του υπάλληλου συναδέλφου και την πρόεδρο για την εξαιρετική επικοδομητική συνεργασία. Και προσβλέπω και μετά τι τερνέ διακοπέ να καταλήξουμε με το καλό από κοινού σε ένα καλό τεκμηριωμένο κείμενο το οποίο θα εκφράζει όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Merci. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Στέβεν, συνεισηγήτρια, για την παρουσίαση αυτή. Θα δώσω αμέσω το λόγο στους διάφορους σκιώδεις εισηγητές. Α, όχι, συγγνώμη, η Μόνικα Χολμάιερ θέλει κάτι να προσθέσει. Ένα μικρό σχόλιο, παρακαλώ. Ναι, παραλίγο να ξεχάσω κάποιον στις ευχαριστίες και θα ήταν ένα φόπα αυτό, στραβοπάτημα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Επίτροπο Τζούλιαν Κίνγκ και όλο του το επιτελείο της Γενικής Διεύθυνσης Home που μας υποστήριξαν και από την ε, Europol, Eurojust, δικαστές εισαγγελείς ήταν πάντα στη διάθεσή μας ώρες ολόκληρες για να μην πω μερόνυχτα ολόκληρα. Όποτε του ζητήσαμε ήταν ε, στο πλευρό μας. Ε, ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Ζίλντε Κέρκοφε που επανειλημμένα ήρθε να μας δώσει υλικό και οι συνεργάτες του. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε Μόνικα Μέγερ για αυτές τις πολύ σημαντικές διευκρινήσεις και δίνω τώρα το λόγο στην Κατερίνα Κινίτσι. Ε, για πέντε λεπτά, αν θέλει. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας, ευχαριστώντας τις δύο συναδέλφους, τη Μόνικα και τη Χέλγα. Και το επιτελείο τους. Καταλαβαίνω όλο ότι επίσης ότι πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσους ευχαρίστησα και εκείνε, εσά, τη γραμματεία, τα επιτελεία όλων των συναδέλφων που συνεργάστηκαν μαζί μας σε αυτή μα ε, την προσπάθεια και τους άλλους θεσμού και οργανισμούς τους οποίους ευχαρίστησαν η Μόνικα και η Χέλγα. Νομίζω πως η εργασία αυτής της Επιτροπής είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει στις θέσεις μας και μέσα στις διαφορετικές μας θέσεις θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι πραγματικά σε ένα κοινό στόχο που είναι πάρα πολύ σημαντικός, δηλαδή η εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών, εξισορροπώντας βέβαια αυτή την ασφάλεια με το σεβασμό των ε, δικαιωμάτων και των ελευθεριών, γιατί αυτού του είδους η εξορρόπηση είναι δυνατή. Να βρούμε ισορροπία ανάμεσα στις δύο αυτές απαιτήσει είναι απαραίτητο και αυτό περιμένουν εξάλλου οι πολίτες από εμά και αυτό ε, επίσης ε, έχει ως εντολή και καθήκον αυτή εδώ η Επιτροπή. Ως προς αυτό λοιπόν ευχαριστώ πραγματικά πραγματικά γιατί εξ αρχής είχαμε μια πολύ αγαστή συνεργασία, σημαντική, που είμαι βεβαία ότι θα συνεχιστεί και θα μας επιτρέψει να φτάσουμε σε αποτελέσματα Πρέπει λοιπόν με αυτή μας τη συνεργασία να είμαστε αποτελεσματικοί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Οι συνάδελφοι έθιξαν ένα σωρό σημεία και βέβαια θα πρέπει να μοιράσουμε το χρόνο μας ανάμεσα σε όλους. Εγώ θα σταθώ σε κάποιες πτυχές, ε, θα δουλέψω με τις τροπολογίες και το πρώτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ε, στο σχέδιο έκθεσης γίνεται καταρχάς μια αξιολόγηση της απειλής και εδώ εντοπίζεται όσο η τρομοκρατία στον οποίο πρέπει εμείς να εμπαθύνουμε. αλλά δεν είναι μόνο ο θρησκευτικός ε, τρομοκρατής η θρησκευτική τρομοκρατία ε, και η Ισλαμική τρομοκρατία. Συμπεριλαμβάνονται εκεί και οι δραστηριότητες ομάδων, μικρών ομάδων, ναι, που είναι εθνικιστές ε, αυτονομιστές, ε, όμως δεν πρέπει να τους ξεχνάμε γιατί και αυτοί χρησιμοποιούν την τρομοκρατία. Ε, και επίσης ε, το έχει υπογραμμίσει και η Ευρωπόλ η οποία υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και αυτής της απειλής. Είναι πολύ σημαντικό και το έχω πει και σε άλλες ε, περιπτώσεις είναι πολύ σημαντική είναι η ανταλλαγή των πληροφοριών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο που είναι διακρατικό και είναι τόσο σοβαρό. Ως προς αυτή την έννοια νομίζω πως είναι σημαντικά όλα όσα έχει υπογραμμίσει η Μόνικα, αλλά θα πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο και να σκεφτούμε και περισσότερο το θέμα της διαλειτουργικότητας για να καταφέρουμε να έχουμε ένα κείμενο ισορροπημένο που θα λαμβάνει υπόψη πάντοτε τα ψηλά στάνταρ ε, ε, όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, αλλά που ωστόσο ταυτόχρονα θα μπορεί να προσφέρει στα κράτη-μέλη μία βάση δεδομένων ευέλικτη ε, και ευλίγιστη ε, για να μπορούν τα κρατημέλη να χρησιμοποιήσουν και ε, τα στοιχεία και να ε, προλάβουν εγκλήματα. Πολύ σημαντική ήταν η ισπανική εμπειρία βέβαια και εδώ θα συμβάλλω και εγώ, αλλά αναμφίβολα είναι μια πτυχή που δικαίως προσέχθηκε πολύ, όπως και το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ευχαριστώ τη Μόνικα που υπογράμμισε ότι εγώ πίεσα για να ενταχθεί και αυτή η πτυχή, επί της οποίας επαναλαμβάνω θα δουλέψουμε κι άλλο. Ένα ακόμα θέμα όπου θα συμβάλλουμε κι άλλο είναι ε, τα μηνύματα πρόθεσης ε, του μίσους η ε, του ε, σε μίσους. Είναι σημαντικό εδώ λοιπόν να τονίζονται τα προπαγανδιστικά αυτά περιεχόμενα, αλλά ταυτόχρονα με αυτές τις δυνατότητες να υπάρχουν και ρεπαρκείς ε, εγγυήσεις σε σχέση με την αφαίρεση του περιεχομένου και να, ώστε να προστατεύεται η ελευθερία έκφρασης. Κάτι άλλο είναι η ροζοσπαστικοποίηση στις φυλακές. Εδώ θα προσπαθήσω να συμβάλλω με μια σειρά από τροπολογίες για να μπορέσουμε να δουλέψουμε λοιπόν στις φυλακές για να μπορέσουμε επίσης να εντοπίσουμε τις πρώτες περιπτώσεις τα πρώτα σημάδια ριζοσπαστικοποίηση και να τα αναχαιτήσουμε. Και πάω γρήγορα γρήγορα στα συμπεράσματα. Σημαντικό είναι ε, το θέμα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ε, το είπε και η Μόνικα και δεν μπορώ παρά να είμαι σύμφωνη. Ε, για το θέμα της διαχείρισης των συνόρων νομίζω πως θα, ίσως θα ήταν χρήσιμο και ευχαριστώ την Προεδρία, τη Γραμματεία και τις συναδέλφους ε, που δέχτηκαν την ιδέα μιας αποστολής στην Ιταλία που νομίζω ακόμα μια φορά έδωσε και την επιβεβαίωση για το πώς δουλεύουμε για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών μέσα στις ευρωπαϊκές χώρες εντάξει, και πιο ιδιαίτερα και στο εξωτερικά σύνορα που τους που είναι η Ιταλική επικράτεια. Είδαμε λίγες περιπτώσεις όπου μπόρεσαν οι τρομοκράτες να διεισδύσουν μέσω των μεταναστευτικών ροών, γιατί δυστυχώς οι περισσότερες ε, τρομοκρατικές απόπειρες έγιναν από ανθρώπους που ήδη ζούσαν στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε λοιπόν να ε, ε, ταυτίσουμε τα δύο θέματα, την τρομοκρατία με τη μετανάστευση. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε την ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα τα εξωτερικά μας. Δηλαδή, ανταλλαγή πληροφοριών, ε, ε, μια ρευστή ανταλλαγή πληροφοριών, μια σωστή κατάρτιση των ανθρώπων που βρίσκονται στα σύνορα για να μπορούν άμεσα να διαπιστώσουν τα μηνύματα των επικίνδυνων ανθρώπων. Στη Σικελία εμείς έχουμε φτιάξει ένα σύστημα που μπορεί μέσω της εμπειρίας και της συμβολής όλων έχουμε φτιάξει ένα σύστημα που μπορεί να εντοπίσει τα πρώτα αμέσως σημάδια. Ίσως θα ήταν ένα μοντέλο λοιπόν που θα μπορούσατε και οι υπόλοιποι να εισάγετε. Ε, είναι πολύ σημαντικό και αυτό γιατί είναι, ε, πρέπει να γίνεται έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα. Και από αυτού πιστεύω πως ε, πρέπει ίσως να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο και δυστυχώς ξεπέρασα το χρόνο που μου δώσατε. Θέλω να, να ευχαριστήσω τις συναδέλφους γιατί ένταξαν ένα θέμα της ε, επιστροφές των οικογενειών των ξένων μαχητών όπως αποκαλούνται, ιδιαίτερα των ανηλίκων γιατί είναι παιδιά τα οποία δυστυχώς γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε εμπόλεμες καταστάσεις και ήδη έχουν ε, ε, ε ίσως στερνιστεί συμπεριφορές πολεμικού τύπου και είναι σωστό να προσεχτούν αυτά τα παιδιά, να στηριχτούν για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα τραύματα αυτά και να ενταχθούν ε, καλύτερα στην κοινωνία. Ζητώ συγγνώμη που ξεπέρασα το χρόνο ε, και σίγουρα θα συνεργαστούμε αγαστά όπως και μέχρι τώρα με τις συγγήτρες και με όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Και τώρα η Μάιτε Παγασαρτοντούα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, ευχαριστίες γνωστές, συμφωνώ και εγώ, ε, για να εξοικονομήσω δευτερόλεπτα, δεν θα τα επαναλάβω. Αυτό το θέμα της τρομοκρατίας έχω, το έχω ζήσει από μια γωνιά της Ευρώπης δεκαετίες ολόκληρες. Γι' αυτό έχω πλήρη επίγνωση τη σημασίας αυτού του εγχειρήματο, αυτού που κάνουμε. Δεν μπορεί κανένα κράτο μέλος μόνο του να κάνει τη δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ. Γιατί εμείς έχουμε μια γενική παρατήρηση, επισκόπηση όλη της κατάστασης και των απειλών και των κινδύνων το τι υπάρχει και το τι χρειάζεται κυρίως να βελτιώσουμε. Σε όλες τις αποστολές που πήγαμε, δικαστές, εισαγγελείς, ε, εμπειρογνώμονες, πρόληψεις μας έχουν ζητήσει πράγματα να κάνουμε από την Ευρώπη. Διότι ακριβώς τα κράτη-μέλη ε, έχουν μια κατάσταση πολύ ετερογενή ως προς την απειλή, ως προς την ιστορία τους, τις δυνατότητες και την ίδια την αντίληψη που έχουν για αυτά τα πράγματα. Άρα το θέμα δεν είναι να αντιμετωπίσουμε μόνο την ε, τζιχατιστική σκοπή τρομοκρατία, αλλά έχουμε και άλλες τρομοκρατίες. Δυστυχώς θα πρέπει να διευρύνουμε ε, τη γωνία ε, υπό την οποία βλέπουμε τα πράγματα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις και μπορεί να συμβουλεύσει κιόλα, σε περίπτωση που δεν έχουμε εμεί την αποκλειστική αρμοδιότητα να συμβουλεύσει πολιτικές για τα κράτη-μέλη που βλέπουν το κάθε ε, ένα από τη δική του μικρή σκοπιά το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το θέμα της τρομοκρατίας είναι διεθνές, υπερεθνικό και θα συνεχίσει να είναι σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Δεν έχει σημασία αν είναι ακροδεξιά, ακροαριστερή τρομοκρατία, ας είναι ό,τι θέλει. Είναι παγκοσμιοποιημένη. Συμφωνώ με την κυρία Κινίτσι για την Ευρωπόλ θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το έργο της, να κάνουμε όσο γίνεται ε, πιο αντικειμενική την ε, περιγραφή. Για τη διαλειτουργικότητα συμφωνούμε όλοι ότι αυτό που χρειαζόμαστε να είναι όσο γίνεται καλύτερα τα στοιχεία και τα δεδομένα, να κάνουμε συστάσεις, να βοηθούν τα κράτη-μέλη, να είναι λιγότερο εγωιστικά, να βάλουν λίγο νερό στο κρασί του τα κράτη-μέλη και να βοηθούν το ένα το άλλο. Θα πρέπει προς τα εκεί να πιέσουμε. Το ίδιο ισχύει και με κάποιους ορισμούς και κάποια ελλείμματα που υπάρχουν και παραθυράκια στα δικαστικά ε, ή στη δίωξη και στο δικαστικό έλεγχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, εκ του νόνου κάνευ, για να υπάρχει ε, εγγύηση ε, για το τι κάνουν τα σώματα ασφαλείας ή διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών. Όλα αυτά υποδικαστικό έλεγχο. Η εμπιστοσύνη βασίζεται στις καλές πρακτικές των κρατών μελών, αλλά και σε ένα σύγχρονο τρόπο αποτελεσματικό ε, αντίληψης για το δικαστικό έλεγχο. Και αυτό δίνει και εγγυήσεις και ε, καθησυχάζει και ανθρώπους που έχουμε διαφορετικές ιδεολογικές αντίληψεις και που προερχόμαστε από διάφορα στρώματα της κοινωνίας. Επτά χρόνια εγώ προσπαθώ στο Κοινοβούλιο και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να τους κάνουν να καταλάβουν, να καταλάβουμε ε, ότι χρειάζονται περισσότερη βοήθεια τα θύματα, να τα ακούμε περισσότερο και να μπορέσουν να επανενταχθούν στην κοινωνία και να τους φερόμαστε καλά, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε καλές προθέσεις αλλά κακές ε, συμπεριφορές. Αυτά. Για τα υπόλοιπα, για την τρομοκρατική απειλή, όπως πολύ καλά είπε η κυρία Κινίτση, το θέμα της μετανάστευσης χρειάζεται διαφορετική μεταχείριση. Δεν είναι στη δική μας αρμοδιότητα. Το κείμενο θα πρέπει να είναι ισόρροπο, ε, αναλογικό. Έχουν κάνει σπουδαία δουλειά οι δύο εισηγητρίες και σίγουρα θα συμπεριλάβουν και πολλές από τις δικές μας προτάσεις για να βρούμε αυτή τη συνοχή και όπου να αισθάνονται άνετα όλες οι πολιτικές ομάδες. Σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης μπορούμε να προχωρήσουμε νομίζω λιγότερο από τη ε, στην ποιότητα των στοιχείων στη διαλειτουργικότητα που είναι δική μας αρμοδιότητα εκκρεμεί αυτό το ζήτημα. Ξέρουμε ότι έχουμε κάνει δουλειά, αλλά θέλουμε ακόμα περισσότερα. Δεν έχουμε φτάσει στο 100% των δυνατοτήτων και των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Υπάρχει κάτι που θα μείνει για το μέλλον και να το σκεφτούμε και αυτό. Συνεργασία, λοιπόν, ανταλλαγή πληροφοριών και όπου υπάρχουν προβλήματα και δεσλειτουργίες θα πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη, να τους βάλουμε ένα καθρέφτη, να δουν τι κάνουν. Ε, να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί για τη χρηματοδότηση της νομοκρατίας. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Είναι κοινέ οι ευθύνε. Αυτό που θα μείνει για το μέλλον ε, έχει να κάνει με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και αυτών των ιδεολογικών φαινομένων. Ευχαριστώ τις δύο συνεισηγήτριες για όλη αυτή τη δουλειά που έκαναν, για όσα προτείνουν και ελπίζω να συμπεριλάβουν και τις δικές μας τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Μάιτε. Πολύ ωραία η σύνθεση αυτή. Η κυρία Ευαζούλη από τους Πρασίνους. Merci Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, θα προσπαθήσω να αντικαταστήσω τον συνάδελφο Γιάννη Φιλίπε που έκανε εξαιρετικό έργο. Ε, είναι δύσκολο να την κατακτηστήσω, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας την κυρία Χορμάγερ και την κυρία Στίβενς για το σχέδιο έκθεσής τους που περιλαμβάνουν, περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία που είναι κλειδιά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εντός Ένωσης. Ιδιαίτερα στηρίζω απόλυτα την μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα κρατημέλη και την περισσότερη ανταλλαγή καλών πρακτικών ε, για την αντίσταση στη, στη ριζοσπαστικοποίηση, προστασία των θυμάτων και καλύτερη τρόπη ε, αντιμετώπισης της χρηματοδότησης της ε, ε, τρομοκρατίας είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικά. Πιστεύω πως μπορούμε να αναπτύξουμε τις περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ε, προσφέρει προστιθέμενη αξία ε, και σκέφτομαι ιδιαίτερα την ιδέα για τη δημιουργία ενώ μιας ευρωπαϊκής μονάδας οικονομικής έρευνας ώστε να μπορούμε να εξετάσουμε καλύτερα τις ύποπτες ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Υπογραμμίζω επίσης ότι είναι σημαντική η περισσότερη και καλύτερη δικαστική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεργασία δεν ε, είναι ποτέ το ίδιο, με, ε, το είναι ένας μόνο επικεφαλής και γι' αυτό και πρέπει να επεκτείνουμε τις αρμοδιότητες του EPO. την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δηλαδή. Ε, νομίζω πως πρέπει να, με, να ρωτήσουμε και να λάβουμε σοβαρά υπόψη όλες τις ειδικέ προτάσεις, ιδιαίτερα να προσέξουμε ε, τα ε, προσωπικά ε, δικαιώματα, δεδομένα, να προσέξουμε πάρα πολύ πριν βάλουμε παντού βιομετρικά στοιχεία. Ξέρετε, εγώ πιστεύω την ανάλυση ε, στοχευμένων στοιχείων και όχι την μαζική συλλογή δεδομένων, πράγμα που είναι πολύ δαπανηρό και επικίνδυνο. Εν γέννη λοιπόν οι συστάσεις πρέπει να ακολουθούν την ιδέα πως μια επιτυχής αντιτρομοκρατική πολιτική δεν σημαίνει ε, σημαίνει μάλλον ε, έναν καθησυχασμό των κοινωνιών που είναι πολύ βασικός, δηλαδή επενδύσεις στην παιδεία, βελτιώσεις στις συνθήκες, στις φυλακές που είναι φρικτές στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως ξέρουμε από την περσινή έκθεση που κάναμε για αυτό το θέμα, ε, και βελτίωση των εξωτερικών μας πολιτικών. Η βασική μου διαφωνία με τον τόνο της ε, έκθεσης είναι ότι η τρομοκρατία παρουσιάζεται ως θρησκευτικό πρόβλημα. Νομίζω πως αυτό είναι σφάλμα. Είναι πολιτικού τύπου βία και δεν μας ενδιαφέρει εάν η έμπνευση είναι ακροδεξιά, ακροαριστερή ή θρησκευτική. Θα πρέπει να αποφύγουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι θεωρούμε πως η τρομοκρατία είναι θρησκευτικό θέμα. Νομίζω πως ε, αυτό εμποδίζει τον περαιτέρω προβληματισμό και μειώνει τον αποτελεσματικότητα του κοινού μας αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Προσβλέπω λοιπόν στις επερχόμενες συζητήσεις τους επόμενους μήνες ώστε να κάνουμε ε, όσο γίνεται πιο χρήσιμες συστάσεις, συνεργασία και να κάνουμε όσα που περισσότερα μπορούμε με βάση τις ακροάσεις και τις μελέτες που έχουμε ήδη κάνει. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η Μαρή Κριστίν Βεριζιά από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τους ε, συγκητές μας, τις συγκητριές μας. Θα ήθελα να μην μακρηγορήσω για να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Με κάποια στοιχεία συμφωνώ. Θα σας παρουσιάσω αυτά τα οποία δεν πολύ συμφωνώ. Γιατί νομίζω ότι δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνουμε αυτά τα, στα οποία συμφωνούμε. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ε, απειλής. Ως περίοδο αναφορά παίρνετε το 1998 μέχρι το 2018. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή την περίοδο παίρνετε ως περίοδο αναφορά, γιατί πολλά έχουν αλλάξει, πολλά έχουν εξελιχθεί μέσα σε αυτή την περίοδο. Να προσέξουμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την περίοδο αναφοράς. Να μην ξεχάσουμε να κάνουμε και συγκρίσεις και με τον αριθμό των επιθέσεων και λαμβάνοντα υπόψη και τι πρόσφατες εξελίξει ε, στην τρομοκρατία και τον αριθμό των θυμάτων. Γιατί οι επιθέσεις θρησκευτικού, ισλαμικού Ισλαμικής ε, ε, φύσης ε, δεν είναι απαραίτητα. Έχουν αυξηθεί, αλλά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία καθολική θεώρηση της τρομοκρατίας και αξιολόγηση της τρομοκρατίας. Θεωρώ ότι επικεντρωνόμαστε κάπως υπερβολικά στο θρησκευτική τρομοκρατία. Δεν λαμβάνουμε υπόψη και άλλες μορφές τρομοκρατίας. Και έχουμε πάντα αναφέρει ότι και οι αποσχετικές στάσεις και οι ακροδεξιές ε, τάσεις και η τρομοκρατία αυξάνονται. Στην ε, Γαλλία έχουμε ένα ακροδεξιό κίνημα το οποίο οργανώνει από ό,τι φαίνεται επιθέσεις. Και λοιπόν η έκθεση θεωρώ ότι επικεντρώνεται κάπως υπερβολικά στην εξωτερική διάσταση της απειλής. Δηλαδή Φυσικά και χρειάζεται να συζητήσουμε και τη διαστασία αυτή, αλλά όπως αναφέρθηκε ήδη, οι πιο πολλές ε, επιθέσεις, ακόμα και ισλαμικές και θρησκευτικέ, ε, δεν ε, διαπράττονται από άτομα από το εξωτερικό της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για μειονότητα. Κοιτώντα λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία που τη διάθεσή μας, και βλέπουμε τις μεταναστευτικές ροές του 2015-2016 έχουμε δύο άτομα από ένα εκατομμύριο. Ε, νομίζω ότι είναι λίγο περαιτή ενέργεια να σπαταλάτε για δύο άτομα από ένα εκατομμύριο. Η υπερβολική επικέντρωση λοιπόν στο θέμα της μετανάστασης πιστεύω ότι υπάρχει φαίνεται ότι αγνοούμε λίγο το, αυτά που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά αυτή τη διάσταση. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δουλειά που έχει γίνει παράλληλα σε ό,τι αφορά τι μεταναστευτικέ ροέ και να μην υπάρχει και αντίθεση με διάφορα θέματα τα οποία επίση απαιτούνται. Το ίδιο ισχύει και για το πακέτο των συνόρων, το Σέγγεν. Και εδώ το Κοινοβούλιο έχει εργαστεί σκληρά και έχει περάσει διάφορα κείμενα. Ο κ. Δεμέρα, από την άλλη πλευρά της αίθουσα, ε, το σύστημα εισόδου-εξόδου θέτει κάποιες αξιώσεις και προϋποθέσεις που αναφέρονται, θα έπρεπε να αναφέρονται εδώ στην ε, έκθεση και σήμερα εγκρίναμε το σύστημα αίτιας, το οποίο επίσης θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει εργαστεί για την διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων. Η έκθεση δίνει την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κάνει τίποτα, δεν εργάζεται για όλα αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν καθολική αποτύπωση όλων αυτών των θεμάτων. Ενδεχομένω να γίνει και μία συνεδρίαση με όλου του συζητητέ που έχουν εργαστεί για όλα αυτά τα θέματα, αλλά μου φαίνεται ότι κάπω εδώ πέρα υπάρχει μία έλλειψη συνεκτικότητα. Συμφωνώ με όλα όσα ακούσαμε για τη συνεργασία των κρατών μελών, μεταξύ κρατών μελών δηλαδή, γιατί πιστεύω ότι αυτό παραμένει ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και η ομάδα Σέγγεν με τον κύριο Κοέλιο εργάζεται για τα θέματα αυτά. Κοιτάξτε λοιπόν τι αξιολογήσει που έχουν γίνει για το σύστημα Σέγγεν και σα διαβεβαιώ ότι είναι δραματικέ. Δραματικό το γεγονό ότι η... υπάρχει τέτοια συμπεριφορά από τα κράτη-μέλη. Άρνηση να μοιραστούν πληροφορίες με άλλα κράτη-μέλη. Κυρία Χολμάιερ. Και κυρία Στίβεντς, δεν θα μείνετε έκπληκτες για το γεγονός ότι θα σας αναφέρω ότι η παράγραφος για τα θεμελιώδη δικαιώματα μου φαίνεται εντελώς ανεπαρκής. Ναι, προφανώς οι πολίτες έχουν δικαίωμα για ασφάλεια. Έχουν δικαίωμα στη ζωή. Έχουν ε, δικαίωμα και στην ασφάλεια. Και προφανώς όλα αυτά είναι θέμα εξισορρόπησης των διαφορών δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει προτεραιότητα σε ό,τι αφορά το ένα ή το άλλο δικαίωμα. Το θέμα είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και να υπάρχει αναλογικότητα. Αυτό επαναλαμβάνεται διαρκώς από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλωστε. Ένα άλλο θέμα δε, το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερος, το ανέφερε αν δεν κάνω λάθος και η κυρία Ευαζολή, το θέμα της ε, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε λοιπόν το θέμα αυτό δεν ξέρω ποιος ε, από τους ομιλητές ε, επέμεινε για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τα εργαλεία τα οποία θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την παρακολούθηση των ατόμων. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία θα έπρεπε πρωτίστως να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της τρομοκρατίας, της, ε, του εμπορίου όπλων, ναρκωτικών και της χρηματοδότησης ε, της τρομοκρατίας. Ακόμα και στο ό,τι αφορά το λαθρεμπόριο έργων τέχνης. Όλα αυτά λοιπόν άλλωστε έχουν και διεθνή παγκόσμιο χαρακτήρα. Πιστεύω δε ότι κάποια στοιχεία τα οποία ζητούνται στην έκθεση θα πρέπει να τα εντάξουμε και στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα όπως το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ήδη έχουν ληφθεί υπόψη διάφορα στοιχεία και θα πρέπει να κοιτάξουμε επίσης το γεγονός ότι η πρόληψη δεν τονίζεται επαρκώς. Άρα η έκθεση συνολικά θεωρώ ότι εστιάζεται προβολικά στις πτυχές της ασφάλειας και όχι επικώς στις πτυχές της πρόληψης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σκέλος της ριζοσπαστικοποίησης. Αν θέλουμε λοιπόν να ε, πετύχουμε κάτι θα πρέπει να εργαστούμε στο επίπεδο των σχολείων, ε, θα πρέπει οι εκπαιδευτές, οι δάσκαλοι να έχουν ιδιαίτερη εκπαίδευση για να εντοπίζουν ε, εγκαίρως τις ενδείξεις και εδώ έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βεριζιά για τις παρατηρήσει αυτές, λέει η Πρόεδρος. Και σε ό,τι αφορά και τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει, ο κύριος Μερτάν δεν είναι εδώ. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην, στον κύριο Μιντή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 10 λεπτάκια. Και αν θα θέλετε να μην υπερβείτε αυτό το χρονικό όριο για να κάνουμε και λίγο καρσιδιάι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε. Δεν θα σχολιάσω την έκθεση ε, και τις λεπτομέρειες της έκθεσης, γιατί αυτό θεωρώ θα το κάνει ο Επίτροπος Κίνγκ που θα έρθει εδώ το Σεπτέμβριο. Είναι τιμή που παρευρίσκομαι σε αυτή την πρώτη συζήτηση του σχεδίου έκθεση. Ιδιαίτερα Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι εδώ, γιατί πιστεύουμε ότι η έκθεση είναι πραγματικά πολύ υψηλή ποιότητα. Από πλευρά δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, πολιτική καταπολέμηση της τρομοκρατία. Νομίζω ότι σε μια πολύ σύντομη χρονική περίοδο καταφέρατε να καταρτήσετε μια αντικειμενική, ισόρροπη έκθεση και αξιολόγηση και πολύ εύστοχη αξιολόγηση του τι έχει ήδη συμβεί για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά επίσης δίνεται και μια φρέσκια εικόνα για το τι συμβαίνει και πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Τι να πρέπει να καλυφθούν και σε ποιους τομείς θα πρέπει να προσαρμόσουμε την προσέγγιση μας. Προτού ακούσω τη συζήτηση, η μοναδική κριτική που είχα ακούσει για την έκθεση αυτή ήταν ότι ενδεχομένω να είναι υπερβολικά μεγάλη σε διάσταση δηλαδή. Αυτό θεωρώ καταρχά ότι είναι θετικό. Αν το μοναδικό που έχουμε να επικρίνουμε για την έκθεση αυτή είναι ότι είναι υπερβολικά μεγάλη, ε, σημαίνει αυτό ότι η ουσία είναι πάρα πολύ καλή. Από αυτά που άκουσα σήμερα το πρωί τώρα. Άκουσα κάποια κριτική. Νομίζω ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ασφάλεια που χρειάζεται μεταξύ ε, ασφάλειας και θεμελιδών δικαιωμάτων, προφανώς η έκθεση ενδεχομένως να μπορούσε να είναι ακόμα πιο σαφής για το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει μια κάποια ισορροπία μεταξύ των δύο πτυχών αυτών. Επίσης, ε, να μην υπάρχει, συμφωνώ, κανένα περιθώριο παρανόησης. Ε, η τρομοκρατία δεν συνδέεται μόνο με τη θρησκεία. Και πραγματικά χαίρομαι που άκουσα δύο παρεμβάσεις από αυτού. Όχι, ούτε είναι κάτι το οποίο συνδέεται με μια εξωτερική και μόνο απειλή. Υπάρχει και εσωτερική απειλή. Και γι' αυτό παρεπιπτόντως ε, είναι τόσο μεγάλο και το τμήμα και το κομμάτι για την ε, καταπολέμηση της ρίζος παστικοποίησης. Επίσης, ε, σας ευχαριστώ που τονίσατε το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχεία φιλοδοξίας και χρηματοδότησης. Προφανώς, πολλές από τις ιδέες θα χρηματοδοτηθούν και τα επόμενα χρόνια. Τώρα, κάποια στοιχεία τα οποία θα ήθελα να τονίσω. Καταρχά, πιστεύω ότι η έκθεση παρουσιάζει με πολύ εύστοχο τρόπο και ξεκάθαρο τρόπο το γεγονός ότι η τρομοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένα θέμα το οποίο το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα πάρα πολύ δυναμικό και σοβαρό παράγοντα ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Αυτό προφανώ όμω δεν υποκαθιστά τι δουλειέ και τι ευθύνε των κρατών μελών. Το τονίζετε πάρα πολύ καλά. Το ότι πρόκειται για κοινή αρμοδιότητα και την αξία των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών που δεν υποκαθιστούν αλλά υποστηρίζουν, συμπληρώνουν τις δράσεις των κρατών μελών. Πρωτίστως όταν καλύπτουμε τις πολλαπλές διαστάσεις ε, της υποστήριξης που δίνουν οι εξωτερικές υπηρεσίες και επίσης ε, την περαιτέρω υποστήριξη που χρειάζεται από τις εξωτερικές ε, ε, υπηρεσίες και από την Europol και από την Eurojust από πλευρά της δικαιοσύνης, από τη Frontex, από τη EULISA σε ό,τι αφορά τα συστήματα πληροφοριών. Μια δεύτερη πτυχή που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι η επικέντρωση η οποία παρατηρείται στην έκθεση στις πτυχές της ε, εφαρμογής. Χαίρομαι που το κάνετε αυτό. Σας ευχαριστώ, γιατί αυτό θα μας υποστηρίξει με τη σειρά του. Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση του επίπεδου υλοποίηση των πολλαπλών αυτών μέτρων που έχουν ε, ανακηρύξει τα τελευταία χρόνια και είναι και μια βασική αρχή την οποία ακολουθούμε σε πολύ σημαντικούς ε, κλάδους όπως είναι η διαλειτουργικότητα. Δεν επικεντρωνόμαστε απαραίτητα στην παροχή νέων συστημάτων, αλλά στην εξέβρεση σωστών τρόπων προκειμένου να αξιοποιήσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο αυτά που ήδη έχουμε, χωρίς να χάσουμε οποιαδήποτε λειτουργία και δυνατότητα έχουμε ήδη αναπτύξει. Για τι πληροφορίε. Και εδώ πιστεύω ότι είναι πολύ ισορροπή η προσέγγιση που ακολουθεί η έκθεση. Αναγνωρίζεται μεν προφανώς η απολύτως απαραίτητη ανάγκη α, να υπάρχουν πληροφορίες, να γίνεται ανάλυση των πληροφοριών αυτών, αλλά και να μοιράζονται μεταξύ των κρατών μελών οι πληροφορίες αυτές. Η αρχή που περιγράφεται στην έκθεση για την κοινή χρήση των πληροφοριών εξορισμού αποτελεί μια σημαντική αρχή. Αν είμαστε λοιπόν, έχουμε ένα κοινό χώρο, αν έχουμε κοινά σύνορα, εξωτερικά σύνορα, είναι προφανές ότι ό,τι πληροφορίες έχει η μία αρχή θα πρέπει αυτόματα να διατίθενται και στις άλλες υπηρεσίες που έχουν ανάλογες ε, υποχρεώσεις προφανώς για την προστασία του κοινού αυτού χώρου. Εδώ θεωρώ ότι έχετε θέσει πολύ σημαντικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την συλλογή των δεδομένων, τη διατήρηση των δεδομένων, τη φύλαξη των δεδομένων. Πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για μα σε ό,τι αφορά και την προετοιμασία των κατευθυντηρίων γραμμών που έχουμε υποσχεθεί. Άρα, διατήρηση των δεδομένων. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, πόσο απαραίτητο είναι να φυλάσσονται τα δεδομένα αυτά για τις έρευνες και για τη δίωξη. Ρίζει σπαστικοποίηση τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ε, εργάζεστε σε αρμονία με την ε, υψηλοπιπέδου ομάδα και που μας δίνεται και περαιτέρω όθηση προκειμένου να ξεπεράσουμε και λίγο τα όρια μας σε ό,τι αφορά το είδος των μέτρων που αναπτύσσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας των ατόμων. Γιατί είναι πάρα πολύ περίπλοκα τα φαινόμενα αυτά. Μιλήσατε επίσης και για την χρηματοδότηση. Εδώ να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερα την κυρία Εύα Ζολή που το είπε τόσο καθαρά και εξάστερα. Υπάρχει σαφής περιορισμός σε αυτά που μπορεί να προσφέρει το τρέχον σύστημα για τη διάθεση χρήσιμων, ωφέλιμων πληροφοριών για την έρευνα και τη δίωξη. Και διαπιστώνουμε τα όρια των όσων πετύχαμε στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ των μονάδων οικονομικής συνεργασία. Και γι' αυτό λοιπόν καταθέσαμε μια πρόταση την οποία και εξετάζεται. Αλλά εδώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πάμε και ακόμα παραπέρα. Θα εξετάσουμε λοιπόν τις προτάσεις σα με πολύ προσοχή. Και το TFTS για να καλύπτονται όλες οι συναλλαγές εφόσον αυτό χρειάζεται. Κρίσιμες υποδομές. Και εδώ. Κάπως ξεχασμένο ήταν το θέμα αυτό. Επικεντρωθήκαμε τόσο πολύ στην κυβερνοασφάλεια που τελικά έμεινε λίγο πίσω το θέμα των κλασικών υποδομών και των κλασικών τρόπων, αν θέλετε, προστασίας των χρήσιμων υποδομών στις κοινωνίες μας. Εδώ όλες οι ιδέες προς συζήτηση θα είναι ωφέλιμες και σε ό,τι αφορά την τρέχουσα αξιολόγησή μας. Ελπίζουμε στο μέλλον και στις μελλοντικέ μας προτάσεις να βρούμε έναν τρόπο για να ανανεώσουμε εκ το τρέχον πλαίσιο που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τέλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, υποσημείωση που βάλατε για την προστασία των θυμάτων. Αναφέρετε όλες τις πτυχές από την εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων μέτρων σε ό,τι αφορά την οδηγία κατά τη τρομοκρατίας, κυρίως, αλλά και τις επιπλέον ιδέες και τα επιπλέον στοιχεία. Αυτό όχι μόνο θα βοηθήσει την κυρία Μίλκε στη δουλειά που κάνει για τα θύματα, αλλά και για μας. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να αναπτύξουμε νέες ιδέες, νέες πρωτοβουλίε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλο προνόμιο για όλους τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας όποτε αυτό χρειάστηκε και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα που πετύχαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν. για αυτή την προσέγγιση και για την ανάλυση. Και τώρα το λόγο μπορείτε να πάρετε και έχω ήδη ε, αρκετούς που το έχουν ήδη ζητήσει. Σας προτείνω να περιορίσετε τις ε, ε, ομιλίες σας στα δύο λεπτά, έτσι ώστε οι δύο συνεισηγήτρες να μπορέσουν να έχουν λίγο περισσότερο χρόνο στο τέλος για να απαντήσουν στις διάφορες ερωτήσεις. Ε, ο κύριος Ντανζόν, καταρχάς, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Δεν θα καθυστερήσω ευχαριστώντα τι εισηγήτριε. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και αυτό ήδη τονίστηκε τους προλαλήσαντες δεν ε, εκφράζομαι ως συντονιστής του ΕΛΚΑ, αλλά εκφράζομαι ε, ε, στο όνομά μου. Είναι προσωπικές μου παρατηρήσεις. Το θετικό είναι ότι όσα είναι τεχνικά είναι πολύ συγκεκριμένα για την διαλειτουργικότητα που κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητη η διατήρηση των δεδομένων γιατί έχουμε πρόβλημα με την με αυτά και φυσικά όσα αφορούν τη χρηματοδότηση αλλά υπόθηκαν ήδη ε, ε, Έχω κάποιες επιφυλάξεις ε, επί του τύπου περισσότερο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια κείμενα που εξηγούμε τη σχέση ανάμεσα στην εγκληματικότητα και την τρομοκρατία. Λες και είναι κάτι καινούριο που μόλις ανακαλύπτουμε και που αυξάνεται διαρκώς. αυτό υπάρχει ανέκαθεν. Τα δίκτυα τα τρομοκρατικά τρέφονται από την εγκληματικότητα προσλαμβάνοντας, ε, στελεχώνοντας τις οργανώσεις τους ε, ε, ε, ξέρουμε εγκληματίες που απλώς μετατράπηκαν σε τζιχαντιστές. Ένα σωρό. Το κείμενα Ωστόσο, ε, κάποιες φορές αναφέρουν δικές μας προσωπικές ε, ε, απόψεις, ενώ οι πυρογνώμονες μας είπαν ότι οι ανταλλαγέ πληροφοριών είναι εντατικές. Υπάρχει, γίνεται, γίνονται ήδη, μπορεί να βελτιωθούν βέβαια, αλλά υπάρχουν. Ναι, η Europal είναι το κατεξοχήν κόμβος μέσω του οποίου θα πρέπει να περνάνε οι πληροφορίες, αλλά εγώ διστάζω κάπως περισσότερο όσον αφορά την αύξηση της Europol σε, όσον αφορά το προσωπικό και τους πόρους, γιατί για μένα οι πόροι και ε, το προσωπικό που δεν είναι και περιόριστο για θέματα τρομοκρατίας θα πρέπει να είναι επιτόπου ε, περισσότερο κοντά στις εθνικές υπηρεσίες που δουλεύουν ε, επιτόπου. Γιατί η Europol δεν έχει νόημα να έχει τεράστιο γραφειοκρατικό όγκο. Ε, πρέπει περισσότερο να, συντονίζω, να συντονίζει. Να είναι ε, ο κατά προτεραιότητα κόμβος όπου θα συγκεντρώνονται και θα διαχέονται τα στοιχεία αλλά όχι να πάρει τεράστιες διαστάσεις. Τώρα για την οργάνωση πρέπει να είμαστε αυστηροί όσον αφορά ε, ε, ενάντια στο Ισλάμ, να κλείσουν ε, η χώρα λατρείας, να διώκονται οι άνθρωποι που κηρύσουν το μίσος και υποστηρίζουν το δρομοκρατία και το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Από την άλλη πλευρά όμως η οργάνωση του μετριοπαθούς Ισλάμ ε, στις κοινωνίες μα είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Εδώ και 30 χρόνια στη Γαλλία το σκεφτόμαστε. Ποτέ δεν τα έχουμε καταφέρει καλά και τέλεια. Εάν βλέπουμε μια δομή που υποτίθεται είναι αξιοσέβαστη και που συγκεντρώνει του μετριοπαθείς και άμεσα μπορεί να παρακαμφθεί από άλλες δομές πιο υπόγειες, πιο κρυφές φυσικά πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι συναρπαστικό θέμα αλλά είναι περίπλοκο ε, στο πλαίσιο των δικών μας εργασιών να δίνουμε οδηγίες για αυτό το θέμα. Ε, ε, είναι πολύ δύσκολο είναι μια ε, θρησκεία που δεν αναγνωρίζει καν ιεραρχίες όπως οι δικές μας θρησκείες με τις οποίες είμαστε πιο εξοικειωμένοι εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Η Άννα Γκόμες. Και εγώ θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τις συζητήτριες και εξάλλου και όλες τη συμβολή των σκιωδών για αυτή τη συζήτηση που νομίζω είναι ε, πράγματα όλα που θα μεταφραστούν στο κείμενο αυτό. Εγώ θα ήθελα από πλευράς μου και βεβαίως... Ε, υπογραμμίζω τα όσα είπε η Κατερίνη και συμφωνώ. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε κάτι που ε, υπογράμμισε και η ΜΑΙΤΕ, ότι χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι μια ευθύνη των κρατών μελών, ναι, μεν, αλλά χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να αναχαιτήσουμε τον διακρατικό, τη διακρατική αυτή απειλή για να ελέγξουμε, για να ανταλλάξουμε πληροφορίες. Αυτό, αυτό πρέπει να επιμείνουμε. Δεύτερον, πιστεύω πως αυτή η έκθεση θα έπρεπε να τοποθετήσει την τρομοκρατία, το φαινόμενο της τρομοκρατίας, μέσα σε ένα ε, παγκόσμιο πλαίσιο. Έχουμε τα στοιχεία της έκθεσης ε, της Europol. Δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι είναι το πιο φρικτό πράγμα που έχει συμβεί και ότι δεν είναι ένα ε, φαινόμενο το οποίο υπήρχε ανέκαθεν. Νομίζω πως αυτή η προοπτική είναι σημαντική. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό το μπέρδεμα και τη σύγχυση που διαρκώς γίνεται απόπειρα να γίνει με την μετανάστευση. Το είπαν και οι συνάδελφοι. Αυτό είναι λάθος και είναι άδικο γιατί είδαμε τι έγινε. Και ό,τι η ιδέα των εκδόσεων είναι λύση. Ε, απελάσεων, συγγνώμη. Ε, Και είπε η Μαρία Χριστίνα ότι δεν είμαστε αρκετά στα θέματα τα κοινωνικά, στην πρόληψη, δεν κάνουμε αρκετά ε, και κατά τη ριζοσπαστικοποίηση ε, τόσο στι φυλακέ όσο και έξω από τι φυλακέ. Και έχει δίκιο. Νομίζω πω αυτό ο τομέα, όπω το είπε και η Κομισιόν αλλά και η Ευαζόλη, η χρηματοδότηση τώρα της τρομοκρατίας θα πρέπει να αναλυθεί καλύτερα και εκεί θα μπορούσαμε να σημάνουμε τη διαφορά γιατί έχουμε δει, μας ρώτησαν μία ε, ε FIU για, την Ένωση το ζητήσαμε για το, για το πλήσιμο ε, του βρώμικου χρήματος. ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ε, μας το αρνήθηκαν εδώ μπορούμε να το βάλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι από τη ΣΥΠΑ Δεν μπορούμε δηλαδή να δίνουμε τα δεδομένα μας, τις είπα και εκείνοι να μην μας τα δίνουν επίσης σε ανταλλαγή. Επίσης έχουμε τα χρήματα που δίνονται στις εγκληματικές ε, οργανώσεις που δίνονται από, από ε, μέσω του συστήματος ΦΠΑ. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έγιναν για ε, το Ισλάμα. Και είναι πολύ σημαντικό να το αν πούμε σωστά γιατί δεν έχει να κάνουμε με τρομοκρατία πραγματικά θρησκευτικού τύπου αλλά πολιτικού τύπου Επίσης ε, απαιτείται και αυτό είναι πολύ σημαντικό η σύνδεση που έχει γίνει με το σχέδιο δράσης CBRN αλλά κατά τη γνώμη μου είναι βάσταχτο τα κάτι μέρη να μην δίνουν πληροφορίες για τις κρίσιμες δομές για τα πυρηνικά. Δεν καταλαβαίνω στην αποστολή που κάναμε να επισκεφθούμε το λιμάνι της Ανβέρσας να μην μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες που μπορούν να μας πούνε τι γίνεται με τους πυρηνικούς που είναι δίπλα στο λιμάνι της Ανβέρσας ε, και χωρίς ε, κάτι τέτοιο αυτή η έκθεση δεν θα έχει νόημα. Είναι ουσιώδες, είναι θεμελιώδες σημασία και είναι πραγματικά ασύλληπτο ότι τα κράτη-μέλη δεν επιτρέπουν να δούμε τι τρέχει εκεί. Συμφωνώ επίσης με τα όσα είπε η Μαρή Κριστίν Περζιά με τις ανάγκες να συνδυαστούμε με τα όσες προσπάθειες γίνονται στη ΛΥΜΠΕ για την διαλειτουργικότητα αν και ήδη περιλαμβάνονται σημαντικές προτάσεις ε, για να μπορέσουμε να ακούσουμε τους διάφορους φορείς επιτόπου. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Σίπελ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αρχίζω με μια γενική παρατήρηση σε ό,τι αφορά την ναι, έκταση της έκθεσης. Γιατί είναι τόσο μακροσκελής. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι θα εντόπιζε τα ελλείμματα και θα έκανε προτάσεις για το πώς θα τα καλύψουμε. Αλλά τώρα η έκθεση αναφέρει θέματα που έχουν λυθεί εδώ και καιρό ή που συζητούνται αυτό τον καιρό. Και διερωτώ με, θέλουμε μια έκθεση που να ονομάζει τα πάντα από την αρχή και να δίνει την εντύπωση ακόμα και στον ε, αναγνώστη που ξέρει τα πράγματα ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα να το σκεφτούμε αυτά τις δομή. Η κυρία Στέβενς μίλησε για την προστασία και τη φύλαξη των συνόρων. Θέλω να τα ξαναπούμε. Η δική μας ε, πολιτική ομάδα έλεγε να έκαθεν ότι τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών είναι ευρωπαϊκά σύνορα και θα πρέπει να φυλάσσονται και να ελέγχονται από κοινού. Εγώ δεν θέλω να χαρακωθούμε και να απομονωθούμε από όλου και πρόσφυγες να μην αφήνουμε. Και όταν πρόκειται για την τρομοκρατία θέλω να πω τα εξή δύο. Η συνάδελφος Κινίτσι τα είπε προηγουμένω ότι Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπόλ, ε, η πλειονότητα των επιθέσεων πέρυσι δεν έγιναν από Ισλαμιστές, τρομοκράτες, αλλά από αυτονομιστές, εθνικιστές και εξτρεμιστές. Από ανθρώπους που ζουν στην Ευρώπη έτσι και αλλιώς και θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας για να ε, παίρνουμε τα σωστά μέτρα και ακόμα και εκεί που συμμετείχαν πρώην πρόσφυγες πολύ συχνά αποδεικνύεται σε λεπτομέρειες ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ρίζος παστικοποιηθεί μετά την έλευσή τους στην Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Κατανοώ αυτά που λέει η συνάδελφος Μόνικα Χούλμαγερ για την υποστήριξη και βοήθεια των θυμάτων. Ωστόσο, ανησυχώ λίγο ταυτόχρονα. Γιατί? δεν είναι τα θύματα των ε, εγκλημάτων ε, θύματα ε, της ομοκρατίας ή των εγκλημάτων είναι θύματα επειδή κάπου βρισκόντουσαν τυχαία. Όλα τα θύματα τα παθαίνουν αυτά τυχαία. Δεν είναι ότι τσακώνονται με την οικογένειά τους και σκοτώνονται. Είναι ότι βρίσκονται εκεί και δεν του νοιάζει το θύμα αν ήταν ε, ληστεία σε τράπεζα ή τρομοκρατική ενέργεια αυτό που του συνέβη. Βεβαίω και θα πρέπει να τους βοηθούμε και να μην τους αφήνουμε στη μοίρα τους. Συμφωνώ επίσης με τη συνάδελφο Χολμάιερ ότι μπορεί ενδεχομένω να υπάρχει ένας λόγος ε, γιατί μάλλον ε, μία από τις αιτίες είναι ε, η Ισλαμιστική τρομοκρατία δεν είναι μονομερής η αντιμετώπιση, δεν νομίζω να το εννοεί έτσι η συνάδελφος, ε, αλλά τώρα έχουμε πολύ συναισθηματικές αντιδράσεις και πολύ φορτισμένη συζήτηση για την τρομοκρατία που συνδέουν με κάποιοι με την μετανάστευση. Προσοχή να κάνουμε τις σωστές συζητήσεις. Για τη διαλειτουργικότητα είπα και προηγουμένως ότι το συζητούμε ήδη και τώρα δεν κατάλαβα τι δουλειά έχει σε αυτή την έκθεση και πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθεί. Αυτόματη ανταλλαγή ε, δεδομένων. Το πρόβλημα δεν είναι καν ότι τα κράτη είναι τόσο απρόθυμα. Αλλά επανέρχομαι σε αυτό που είπε προηγουμένως ο συνάδελφος Ντονζό. Πολύ συχνά οι διοκτικές μας αρχές, ε, οι αστυνομίες δεν έχουν το προσωπικό και δεν έχουν και την υλικοτεχνική ε, υποδομή, γιατί είναι και διαφορετικός ο ορισμός για τη βαριά αξιόπινη πράξη και για την τρομοκρατική ενέργεια. Δηλαδή τι θα ανταλλάσσουν, ούτε για αυτό δεν συμφωνούν. Και επίσης υπάρχει και ασάφεια για την ποιότητα των δεδομένων, όχι μόνο η τεχνική, δηλαδή πώς παίρνεις αποτυπώματα και αν είναι αξιόπιστο αυτό, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή από πότε Ε, ένα στοιχείο, μια ένδειξη είναι τόσο, η αναγνώριση κάποιου στοιχείου είναι τόσο αξιόπιστη ώστε να μπει σε μια τράπεζα δεδομένων. Είπε ο ο Σκίνγκο Επίτροπο ότι χρειάζεται διευκρίνηση για να μην κάνουμε κανένα λάθο. Και το τελευταίο για τα κηρύγματα μίσου και τη διάδοση. Δεν ξέρω αν το σωστό μέτρο είναι απάλληψη περιεχομένου από το ίντερνετ και λόγω του ρατσισμού, του εθνικισμού και ε, της μυσαλλοδοξίας θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη δημοκρατία και όχι να σβήνουμε ότι δεν μας αρέσει ή μπορεί να είναι επικίνδυνο. Δεν λύνει αυτό τίποτα. Χρειάζεται να αντιπαρατεθούμε με αυτά τα πράγματα για να είναι ο κόσμος ε, ενήμερος και να μην τρέχει πίσω από αυτά τα ε, κηρύγματα τυφλός και ο ίδιος. Ευχαριστώ για τα σχόλια αυτά κυρία Ζίπελ. Θα απαντήσουν οι συνεισηγήτρες φαντάζομαι, μια πρώτη απάντηση θα δώσουν και θα δοθεί και συνέχεια στους επόμενους μήνες. Ο κύριος Φρουνζουλίκα για δύο λεπτά. Δύο εσείς, δύο, δύο. Ε, Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και θα ήθελα να σας ζητήσω εφόσον γίνεται να καταρτιστούν οι τροπολογίες σε μία γλώσσα, γιατί αν θα γίνουν οι τροπολογίες σε όλες τις γλώσσες, Έκλεισε το μικρόφωνο του μιλητή. <laughs> Να γίνουν λοιπόν οι τροπολογίε σε μία γλώσσα. Γιατί αν γίνουν σε όλε τι γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρεθούμε σε φρικτή κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν, γιατί μια και μιλάμε πολύ γαλλικά, να το πούμε, κάνουμε στα γαλλικά τι τροπολογίε. Γιατί μιλάμε για διαφορετικού όρου. Όρου διαφορετικού σε διαφορετικέ γλώσσε. Uh, Για την έκθεση που παρουσιάστηκε λοιπόν τώρα. Νομίζω ότι η έκθεση δεν ε, τονίζει επαρκώς κάποιες σημαντικές πτυχές. Επιτρέψτε μου να ε, αναφέρω κάποιες εξ αυτών. Η έκθεση δεν αναφέρει, δεν τονίζει το ασθενές σύστημα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, ασθενείς και μη συντονισμένη εφαρμογή των, εθνικ... των ε, συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατακαιρματισμένες βάσεις δεδομένων. Ανεπαρκείς, έχουμε πάρα πολλές βάσεις δεδομένων. Δέκα και παραπάνω που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό και γίνεται χαμός. Περιορισμένη πόρη και υποστήριξη των δυνάμεων ασφαλείας σε κάποια κράτη-μέλη. Δεν θέλω να το αναφέρω ονομαστικά, αλλά κοιτώντα ε, τη χρηματοδότηση για τις ε, δυνάμεις ασφαλείας, τις δυνάμεις κατά της τρομοκρατίας, τις ειδικά σώματα, υπάρχουν χώρες που αφιερώνουν πολύ χαμηλό προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό. Και ξέρετε ότι οι τρομοκράτε τι έχουν μελετήσει επακριβώ αυτέ τι καταστάσει και τι εκμεταλλεύονται. Επίση, τεράστια προβλήματα σε διαφορά αφορά τι μυστικέ υπηρεσίε, μεγάλε αποτυχίε και γι' αυτό έγιναν όλε αυτέ οι τρομοκρατικέ επιθέσει μέσα στην καρδιά τη Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την εποπτεία, την ανείχνευση, την προτεραιοποίηση, ε, την ιεράρχηση των απειλών και σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα στα δεδομένα. Όλα αυτά θα πρέπει να αναφερθούν γιατί αυτή η έκταση θα τύχει ανάλυση από όλες τις δυνάμεις ασφαλείας, τα Υπουργεία Ιστορικών, Εξωτερικών, Άμυνας, τις μυστικές υπηρεσίες όλων των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να χορηγήσουμε μια συνεχτική και πλήρη έκθεση. Επίσης, προβλήματα με τα δικαστικά συστήματα δεν τονίζονται παρκώς. Υπάρχουν διαφορές και στους νόμους και στην ε, νοοτροπία και την κουλτούρα και την ασφάλεια. Για παράδειγμα, πολύ σύντομε φυλακίσεις ε, των ε, εγκληματιών που έχουν διαπράξει επιθέσεις τρομοκρατικές. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό σύστημα σε ό,τι αφορά την κατάσταση αυτή. αναφέρθηκε. Μεν θα πρέπει να τονιστεί πιο πολύ. Όμως, γιατί έχουμε χαμηλά αποτελέσματα, πολύ απογοητευτικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τη ριζοσπαστικοποίηση. Άρα, ανεπαρκή πόροι και σε πολλές περιπτώσεις έλλειψη της λογοδοσίας σε ό,τι αφορά τις μυστικές υπηρεσίες στην αστυνομία και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Επίσης, χαμηλή πόρη σε ό,τι αφορά τις τεχνικές ε, διαστάσει, τεχνική διάσταση των τεχνικών πόρων. Έλλειψη πλήρους εφαρμογής, ε, ανεπαρκής εφαρμογή των ε, βασικών εργαλείων όπως το PNR, όπως το πλαίσιο πριν, το σύστημα για τις θεωρήσεις, φρεχτή κατάσταση. Πώς γίνεται, να μην είναι καν διασυνδεδεμένα αυτά τα συστήματα, αυτές οι βάσεις δεδομένων. Πρέπει κανείς να κάτσει να τα εξετάσει ένα προς ένα. Πρέπει όλα τους αυτά να είναι διαλειτουργικά, να είναι διασυνδεδεμένα. Και θα πρέπει να αναφερθεί πιο πολύ το γεγονό ότι υπάρχει αύξηση του λαθρεμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εδώ ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση των ε, των τρομακτικών δικτύων προέρχεται από απάτες, από ληστείες, από λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών, από εγκλήματα και τέλος η διαφορετική προσέγγιση μεταξύ κρατών μελών. Πώς να εφαρμοστούν όλα αυτά όταν δύο χώρες τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τέτοιο ρόλο δεν είναι ακόμα στο χώρο Σέγγεν, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Πώς είναι δυνατόν, πώς να λειτουργήσει αυτό το σύστημα όταν μπαίνει ο κόσμος χωρίς πρόβλημα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε καλύτερα λοιπόν τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και για να ολοκληρώσουμε το ΚΑΤΣΔΙ η Ελένα Βαλενθιάνο. Αν θέλει να τηρήσει το δίλεπτο. Ε, Βεβαίω. Euh, Μάλιστα έχουν υποθεί σχεδόν όλα και με έχουν καλύψει από αυτά που θα έλεγα εγώ. Και συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Κινίτση, η κυρία Βερζιά και οι Αναγκόμες και λοιποί και ο κύριος Ντανζάν. Ε, το μόνο πρόβλημα που βλέπω εγώ από την έκθεση ε, που βεβαίως πάντα χωράει βελτιώσεις με τη βοήθεια όλων των συναδελφών είναι ότι υπάρχει ένα ιδεολογικό στίγμα εδώ πέρα στην έκθεση και έχει σχέση με το Ισλάμ. Δηλαδή, αν πρέπει να ορίσουμε τι έστι ριζοσπαστικό Ισλάμ και ακραίο μεταξύ μας, δεν θα συμφωνήσουμε. Τουλάχιστον στα ισπανικά η λέξη «radical» δεν είναι βρισιά ραντικάλ είναι κάτι ριζικό, ριζοσπαστικό που πάει στη ρίζα των προβλημάτων. Άλλο το ε, ε, ακραίο Ισλάμ και άλλο το βίο Ισλάμ ή το εξτρεμιστικό και άλλο το ριζοσπαστικό ε, που, που, που ενέχει προθέσεις ε, βίας. Δεν είναι ο ίδιος ο λόγος μίσους και το κήρυγμα του ριζοσπαστικού Ισλαμισμού. Λοιπόν, Ισλάμ, συγγνώμη. Και τι λέμε λοιπόν, ότι καλούμε τα κράτη-μέλη να ανέχονται μόνο τις πρακτικές του Ισλάμ εντός εισαγωγικών που συνάδουν πλήρως με τις αξίες της Ένωσης. Μα τι στο καλό σημαίνει αυτό το πράγμα. και σαβεντήρ. Και ποιες είναι οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να επιτρέψουν κάποιες πρακτικές στο Ισλάμ. Για το κείμενο που έχω μιλάω, σε ισπανικά το έχω. Είναι το μόνο που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να εξηγήσω την κατάσταση. Λοιπόν, για μένα ε, είναι, το πρόβλημα είναι αυτή η θεωρητικοποίηση που κάνει η έκθεση για το Ισλάμ. Γιατί όλα αυτά τα τεχνικά και συστάσεις που μπορούν να βελτιωθούν, που ήδη υπόθηκαν, όπως είπε και η κυρία Κινίτση και τα λοιπά, δεν με ενοχλούν τόσο πολύ. Αυτό που με ανισχύει είναι ότι ορίζουμε εμεί τι είναι ριζοσπαστικό Ισλάμ και ποιε πρακτικές μπορούν να συνάδουν με τις αξίες της Ένωσης και ποιε είναι αυτές. Να πάνε να πνιγούν δηλαδή μετανάστες, αυτές είναι οι αρχές ε, γιατί αυτή τη στιγμή, μη τι άλλο, αμφισβητούνται οι αξίες της Ένωσης. Όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το Ισλάμ και τη μετανάστευση κλπ. Ε, χρειάζονται χοντρό έλεγχο. Συνενετικό, εντάξει. Γιατί τουλάχιστον εγώ δεν διαφωνώ. Και ε, αυτά που λέει η έκθεση για τον ορισμό για το τι είναι κρέο Ισλάμ και όχι και τι θα κάνουμε τους μετριοπαθείς όπως είπε ο Ντανζάν εμείς θα ορίσουμε ποιοι είναι μετριοπαθείς και θα τους κάνουμε. Όλο αυτό ε, μου φαίνεται ένα σύνοθήλευμα έτσι πάρα πολύ αμφισβητούμενο και συζητήσιμο. Εκτό από τι τροπολογίε για το υπόλοιπο και τι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδες να το συζητήσουμε. Βεβαίω, κατά τα άλλα ευχαριστώ πάρα πολύ για την καταπληκτική δουλειά και τις προσπάθειέ σα. Ευχαριστώ πολύ Ελένα και για αυτή την ταχύτητα. που εντοπίσατε τα θέματα που χρειάζονται δουλειά το επόμενο διάστημα. Παρ' όλα αυτά θα δώσω φυσικά το λόγο στις δύο συνεισηγήτρες. Ε, μοιραστείτε το χρόνο που μας ε, απομένει και πιο γρήγορα αν θέλετε να τα πείτε. Ε, αλλά στις 11 τελειώνουμε. Και από εδώ και πέρα αρχίζει η επόμενη προσπάθεια για το σχέδιο έκθεσης με τροπολογίες κλπ. Δεν ξέρω με ποια σειρά θέλετε. Με τη σειρά που θέλετε. Πρώτη Χέλγα και μετά η Μόνικα γιατί το κάναμε προηγουμένως με την αντίστροφη σειρά. Όπως θέλετε. Alors, Έχει Έλγα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ειλικρινά ε, για την ε, επικοδομητική στάση σας. Προσπάθησα να σας ακούσω όλους, ε, σημειώσαμε τις ε, παρατηρήσεις. Χρόνο δεν έχουμε φυσικά αρκετό για να απαντήσουμε τώρα όλες τις παρατηρήσεις. Θα τα ξαναδούμε μετά τις διακοπές. Σίγουρα θα τα συζητήσουμε από κοινού. Σε κάθε περίπτωση περιμένω τις τροπολογίες σας και με βάση αυτές θα μπορέσουμε στη συνέχεια να βελτιώσουμε το κείμενό μας. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποια σχόλια και τώρα σε σχέση με το Ισλάμ από τον κύριο Βαλενθιάνο ε, ε, καταλαβαίνω αυτά που λέει. Ε, να το κοιτάξουμε από κοινού πώς μπορούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Εγώ νομίζω ότι με τη Μόνικα προσπαθήσαμε να έχουμε μια καλή ισορροπία και για το Ισλάμα. Αν θεωρείτε ότι είναι κάπως ανεπαρκή αυτά και θέλετε να κάνετε προτάσεις, τις καλωσορίζω και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το κείμενο. Σε ό,τι αφορά τη σχέση κρατών μελών και ευρωπαϊκού επίπεδου, συμφωνώ απολύτως ότι τα θέματα τα επιχειρησιακά θα πρέπει να βρίσκονται στα χέρια των κρατών μελών και η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί θα πρέπει κυρίως να επικεντρώνονται στην υποστήριξη και στη διευκόλυνση της δράσης ε, των κρατών μελών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτή είναι η αισθήση δική μας. Η Europol που ήδη τώρα υποστηρίζει τις εθνικές αρχές και τις αστυνομικές αρχές στην αστυνομική έρευνα και στη δίωξη. Ε, προφανώς το κάνει τώρα και αυτό θα συνεχίσει να κάνει και δεν θα υποκαθιστά ε, τις εθνικές αρχές. Παίζει σημαντικό ρόλο η Europol στην αποκρυπτογράφηση κάποιων μηνυμάτων γιατί ορισμένα κράτη-μέλη δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Για τα εξωτερικά σύνορα Κατάλαβα τις παρατηρήσεις για τη σύνδεση της τρομοκρατίας με την μετανάστευση. Ε, κατανοώ τις επικρίσεις σας. Εγώ δεν, είπα ποτέ ότι, δεν είπαμε ότι όλοι οι μετανάστες είναι τρομοκράτες. Επίσης είπαμε ότι είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Και βεβαίως ε, δεν θα πρέπει όμως να φλούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται ε, τα μεταναστευτικά ρεύμα, τις ροές αυτές για να εισέρχονται στην Ευρώπη, για να διεισδύουν. Και υπάρχει αυτό. Ο Αμπτελσλάμ μπόρεσε ε, να εκμεταλλευτεί ε, τις μεστατευτικές ροές για να κάνει επιθέσεις ε, στις Βρυξέλλες και στη Γαλλία και πήγαινε ερχόταν κιόλα. Και δεν είναι είτε το ένα είτε το άλλο, είναι και το ένα και το άλλο. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας λοιπόν είναι πάρα πολύ περίπλοκη υπόθεση και εμείς έχουμε να κάνουμε με πολλούς εταίρους εκεί ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό ε, και πρέπει να συνεργαστούμε για να συμπληρωθούν όλα τα κομμάτια του πάζελ και να ε, βγουν όλα στο φως. Και αυτό το πάζελ μαζί θα το συμπληρώσουμε για να έχουμε όλα τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα, να μπορούμε να τα συνδυάσουμε και να τα φέρουμε στη συζήτηση. Θέλουμε να τονίσουμε ότι όλα φυσικά αυτά είναι κρίσιμα και δεν προσπαθούμε να αποκλείσουμε κάτι. να βάλουμε υπόψη και κάποια θέματα που δεν μας αρέσουν πάρα πολύ. Επίσης, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι προς Νότον συνορεύουμε μετά τη Μεσόγειο με τη Λιβύη, που είναι χώρα ε, ξοφλημένη. Failed state. Και το ISIS αλωνίζει στη Λιβύη. Τι θα κάνουμε λοιπόν δεν θα τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει βεβαίω να προστατεύουμε τα νότια σύνορά μας εξωτερικά πάρα πολύ καλά. Επίσης δεν θα πρέπει να λησμονείτε ότι στην ε, Συρία και στο Ιράκ υπάρχουν ακόμα κάποιοι μαχητές που θέλουν να γυρίσουν στην Ευρώπη. Και αυτό μπορεί να γίνει με τη μετανάστευση ή και με την αεροπορία. Πάρουν μια πτήση. Και εκεί θέλει προσοχή για τον επαναπατρισμό των ξένων μαχητών. Σε ό,τι αφορά την ευθύνη, συμφωνώ με όλες τις παρατηρήσεις. Θα πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε να τσακίσουμε την τρομοκρατία. Η ασφάλεια είναι εθνική αρμοδιότητα μεν και θα παραμένει και παραμένει. Τα ξέρουμε αυτά στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουμε άλλη προσέγγιση, ε, τα λένε συνθήκες. Θα πρέπει να καλέσουμε όλα τα κράτη-μέλη για να συνεργαστούν καλά και να υπάρχει ασφάλεια ε, να προέχει προς όφελος όλων. Και υπάρχει και προστιθέμενη αξία για όλους έτσι ώστε να εγγυόμαστε την ασφάλεια αλλά και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Θέλουμε να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή. Και πάλι εδώ δεν είναι ή το ένα ή το άλλο και τα δύο. Τέλος, ευχαριστώ όλους. Περιμένω τις τροπολογίες σας και θα συνεχιστεί η συζήτηση μετά τις ενές διακοπές. Σταματήσω εδώ να μιλήσει λίγο και η κυρία Χόλμαγερ. Σας ευχαριστώ, Μονικά. Πέντε λεπτάκια έχετε. Και να σα υπενθυμίσω, αν ε, φύγουν όλοι τελευταία στιγμή, είναι ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών μετά από αυτά που μας είπε η κυρία στιβεν είναι 11 Σεπτεμβρίου και ε, συμβολική ημερομηνία 12 το μεσημέρι. Μόνικα, 5 λεπτάκια. Ευχαριστώ πολύ Ναταλή. Και καταρχάς, στο θέμα της ριζοσπαστικοποίηση. δεν είχε κάνει τόσο πολύ ε, εντύπωση ως τώρα, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι ε, εννοώ με τα μέτρα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, οποιασδήποτε μορφής ριζοσπαστικοποίησης, αριστερής, δεξιάς, ρισκευστικής, ό,τι ριζοσπαστικοποίησης θέλετε. Κάθε μορφή ε, ρίζοσπαστικοποίηση και εξτρεμισμού θα πρέπει να καταπολεμάται και γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται κοινωνικά μέτρα. Οι παρατηρήσεις σου φυσικά είναι δικαιολογημένε και σωστέ. Το πρόβλημα είναι ότι όντω ω τώρα δεν είχαμε επαρκή εμπειρογνωμοσύνη σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπάθησα πραγματικά να ψάξω. Υπάρχουν πολλέ ΜΚΟ, υπάρχουν κάποιε ακαδημαϊκέ έδρε οι οποίε δεν συνεργάζονται και δεν μεταβιβάζουν αυτή τη γνώση που έχουν. Και άρα η βασική σκέψη είναι η εξή. Ανεξαρτήτως για τι μορφή ριζοσπαστικοποίηση και εξτρεμισμό μιλάμε, ανεξάρτητα από τα αίτια που έχει προκύψει, θα πρέπει να μαζέψουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, όλη αυτή τη γνώση. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν και να δημιουργήσουμε κέντρα αριστείας κατά της ριζοσπαστικοποίηση, κατά του εξτραμισμού, προκειμένου το επιστημονικό αυτό έργο, το οποίο ως τώρα προερχόταν από τοπικά πολύ καλά προγράμματα ένταξης, ενσωμάτησης, καταπολέμησης ριζοσπαστικών τάσεων και εξελίξεων σε διάφορες περιοχές. Όλα αυτά λοιπόν, όλους αυτούς ο όγκους πληροφοριών να συγκεντρωθεί σε ένα σημείο. Είναι και θέμα χρηματοδότησης προκειμένου να υπάρχει τέτοια ανταλλαγή. Αλλά δεν υπάρχει πραγματικά κάποια εμπειρογνωμοσύνη, αριστεία, με συντονισμένο τρόπο να λειτουργεί. Και να είναι και στη διάθεση των ε, πολιτικών ευθυνόντων. Ακόμα και η επιλογή των ε, όρων στα διάφορα επιστημονικά κείμενα δεν εμ, είναι συνεκτική και είναι μεγάλες διαφορές, μεγάλες διαφορές ακόμα και μεταξύ των εμπειρογνωμόνων σε ό,τι αφορά τη ριζοσπαστικοποίηση, τον εξτρεμισμό και σε ό,τι αφορά το Ισλάμ. Δεν είναι. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μέτριο οι Ισλαμικές, ε, μουσουλμανικές οργανώσεις που τηρούν τις ε, αρχές και τις αξίες ε, του χάρτη ανθρωπινών δικαιωμάτων. Και θα ήθελα να τονίσω ότι οι εξτρεμιστές δεν υποστηρίζουν και δεν συνάδουν με τον χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων και να ευχαριστήσουμε αυτούς που το κάνουν. Τη μουσουλμανική λοιπόν κοινότητα που καταβάλει την προσπάθεια αυτή για συνεργασία, για ένταξη, ενσωμάτωση, για το συντονισμό με τις διάφορες αρχές. Το καλωσορίζουμε αυτό. Δεν ε, θέλω λοιπόν να κάνω εικασίες, αλλά ε, αναφέρονται και κατευθυντηρίε γραμμές σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την εκπαίδευση των μημάμιδών κατά πόσον υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπως στην Ιταλία και η Γερμανία έχει δύο-τρία πανεπιστήμια και στη Γαλλία γίνονται κάποιες απόπειρε ε, για να υποστηριχθεί όλη αυτή η διαδικασία προκειμένου στην Ευρώπη και σε πανεπιστημιακό επίπεδο να υπάρχει σωστή εκπαίδευση. Αυτό είναι θετικό, χωρίς φυσικά να προδιαθέτω το περιεχόμενο. Das Wesentliche ist, dass uns aber die Experten hier auch eines sehr klar gesagt haben. Das möchte ich sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Αυτό λοιπόν θέλω να το εκφράσω με πάσα σαφήνεια, ότι υπάρχουν εξτρεμιστές, ε, Ισλαμιστές που χρησιμοποιούν μόνο ένα 4% του Κορανίου. Αυτό λοιπόν μας το ανέφεραν διάφοροι εμπειρογνώμονες. Αυτούς δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να λονίζουν και να διακηρύσουν τις ιδέες τους. Ανακοίνωση των διερμηνέων. Εδώ σταματάει η διερμηνία σύμφωνα με την προηγούμενη ανακοίνωση γιατί είναι η 31η μέρα της απεργίας μας ε, και είπαμε ότι θα σταματήσει η διερμηνία στις 11. Σε ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.